Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε στο πρόγραμμά μας ανταλλαγή απόψε με τον Άντερ Φόγκ Ρασμούσεν, Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, με θέμα το μέλλον της Ευρωπαϊκής Άμυνας. Μια προοπτική του ΝΑΤΟ. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον Γενικό Γραμματέα Ράσμουσεν σε αυτή την κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής μας με την Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας και επίσης θα ήθελα να καλωσορίσω τους συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια από έξι χώρες. Πάει ένας χρόνος από τότε που είχαμε τελευταία συνάντηση με ε, τον κύριο Ράσμουσεν επ' ευκαιρία της ε, διάσκεψης κορυφής του Σικάγο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον ΝΑΤΟ επίκαιρη αυτή η συνάντηση, γιατί το ΝΑΤΟ αντιμετωπίζει ε, και η Ευρωπαϊκή Ένωση σημαντικές ε, προκλήσεις με το Αφγανιστάν, Ιράν, Συρία και εν ώψη και του Συμβουλίου Κορυφής του Δεκεμβρίου. Αυτά τα δύο θέματα, επιχειρησιακές προκλήσεις και σε θέματα Σομαλίας, ε, Σαχέλ και η ανάγκη βελτίωσης ε, της ε, αμυντικής μας συνεργασίας στην Ευρώπη είναι κρίσιμα θέματα. Μάλιστα, τη στιγμή μιας οικονομικής κρίσης και πολιτικής αβεβαιότητας. Ήθελα να υπενθυμίσω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιχειρηματολογούσε ε, έμανα ως προς τη συμπληρωματικότητα του ΝΑΤΟ με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την Ευρωπαϊκή Τετραντική και την παγκόσμια ασφάλεια. Και μάλιστα η συνθήκη της Λισαβόνας επιβεβαιώνει το ζωτικό ρόλο και των δύο μερών. Είναι σημαντικό λοιπόν στις διακηρύξεις ε, ε, και στη συνθήκη να επενδύσουμε στην αμυντική συνεργασία πριν η λιτότητα και οι περικοπές υπονομεύσουν την δυνατότητά μας να φροντίσουμε για την ασφάλειά μας και στην κοντινή και στην γειτονία μας. Και μάλιστα το Δεκέμβριο το Συμβούλιο Κορυφής ε, θα έχει μια μοναδική ευκαιρία για να ε, επεξεργαστεί τη δυνατότητα βαθύτερης και ευρύτερης αμυντικής συνεργασίας, βελτιώνοντας ε, τις διάφορες ε, δομές συνεργασίας, μόνιμες και άτυπες, και η καλύτερη χρήση της συνεργασίας αυτής, καθώς και τη χρήση των ομάδων των μάχημων ομάδων. Και επίσης θέλουμε σημαντικές συνεργασίες και σύσφυξη των συνεργασιών όπως αυτής με τον ΝΑΤΟ. Θα ήθελα να εκφράσω την ανησυχία μου για την κλιμάκωση των επιθέσεων στο Αφγανιστάν, να και μπήκαμε σε μάχημη περίοδο και μάλιστα είδαμε πόσες ζωές χάθηκαν. Την περασμένη εβδομάδα 7 στρατιώτες του ΝΑΤΟ έχασαν τη ζωή τους εκεί. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς πιστεύετε θα εξελιχθεί η κατάσταση της ασφάλειας ε, μετά την αποχώρηση των στρατευμάτων της ΑΕΣΑΠ. Λοιπόν, θα θα σταματήσω εδώ και θα δώσω σε εσά το λόγο για την παρουσίαση. Παρακαλώ, έχετε το λόγο κύριε Ράσμουσεν. Thank you very much, Mr. Provera, for that. Σας ευχαριστώ κύριε Προβέρα για την ευγενική σας εισαγωγή. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι και πάλι εδώ και συναντιόμαι με τα μέλη των δύο επιτροπών και με τους συμμετέχοντες ε, στα Εθνικά Κοινοβούλια στι αντίστοιχε επιτροπέ, στα μέλη των επιτροπών. Τακτικά συναντιόμαστε και χαίρομαι λοιπόν που βλέπω πολλά οικία πρόσωπα. Προσβλέπω λοιπόν σε άλλη μία ζωντανή συζήτηση. Θα ήθελα λοιπόν να σημειώσω καταρχάς κάποια στοιχεία. Είμαι απόλυτα δεσμευμένος για μια ισχυρή και ανοιχτή Ευρώπη και πιστεύω κράταντα ότι η Ευρώπη θα πρέπει να έχει μια ισχυρή κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας. Χαίρομαι που θα υπάρξει, θα γίνει ειδικό συμβούλιο, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, για τα θέματα ασφάλειας και άμυνας τον επόμενο Δεκέμβριο. Θα είναι η πρώτη φορά ουσιαστικά από την αρχή της διεθνούς δημοσιονομικής κρίσης που οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα επικεντρωθούν σε αυτή την σημαντική πτυχή μια ισχυρή και ενωμένη Ευρώπη. Θα ήθελα ωστόσο να είμαι και ειλικρινή. Αν τα ευρωπαϊκά έθνη δεν δεσμευτούν σταθερά σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις στον κλάδο της άμυνας και της ασφάλειας, όλα τα λόγια για την ισχυρή πολιτική, για την άμυνα και την ε, ασφάλεια θα είναι κενά, άδεια. Και δεν πρόκειται να μας βοηθήσει να προσεγγίσουμε την ισχυρή Ευρώπη, την Ενωμένη Ευρώπη που όλοι θέλουμε. Κοιτώντα λοιπόν το μέλλον, ατενίζοντα το... τι προοπτικέ μέχρι το Δεκέμβριο, θα πρέπει τρία πράγματα να έχουμε στο μυαλό μα. Καταρχά, εμεί οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι μόνο τα μέτρα ήπιας δύναμης είναι ανίσχυρα χωρίς πραγματικές ικανότητες οι οποίες θα υποστηλώσουν τη διπλωματία της η, Ευρωπαίοι, η Ευρώπη δεν θα έχει καμία επιρροή και καμία αξιοπιστία. Θα διακινδυνεύσει να μείνει θεατής των παγκόσμιων τεκθενόμενων παρά ο ισχυρός φορέας που θα μπορούσε και θα έπρεπε να είναι ο ισχύρο παράγοντα που θα έπρεπε να είναι. Η εμπειρία μας στα Δυτικά Βαλκάνια καταδεικνύει αυτό ακριβώ. Η σταθερότητα και η, ε, η επανάκτηση της σταθερότητας προαπέτησε ένα μείγμα ήπιας και πραγματικής ε, δύναμης και το είδαμε αυτό σε ό,τι αφορά την συμφωνία την πρόσφατη μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινα. Η η συμφωνία αυτή έγινε μετά από τη μεσολόβηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγχαίρω τον κάθε άστον για την εξαιρετική της δουλειά. Αλλά και οι δύο πλευρές ήθελαν το ΝΑΤΟ να διαβεβαιώσει ότι θα υπήρχε η απαραίτητη ασφάλεια για την εφαρμογή της συμφωνίας. Κατά δεύτερον, η μείωση της ευρωπαϊκής άμυνας και η περικοπή των σχετικών δαπανών αναπόφευκτα θα μας οδηγήσει σε περιορισμένο ρόλο της Υπήρου μας στο διεθνές προσκήνιο. Η Ευρώπη δεν θα είναι σε θέση να συμμετάσχει στην διαχείριση των κρίσεων. Ο μοναδικός τρόπος αυτό να αποφευχθεί είναι να σταματήσουν οι περικοπές σε ό,τι αφορά τις, την άμυνα και να υπάρξει νέα επένδυση στην ε, ασφάλεια μόλις ανακάμψουν οι οικονομίες μας. Εν τω μεταξύ, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε με καλύτερο τρόπο, να αξιοποιήσουμε με καλύτερο τρόπο αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας για να ενεργήσουμε από κοινού ως Ευρωπαίοι στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του ΝΑΤΟ για να μπορέσουμε να έχουμε τις πολύ ακριβές ε, υποδομέ ασφάλειας που δεν μπορεί καμία χώρα να πληρώσει από μόνη τη Τέλος. Είναι σημαντικό να, υπάρχουν, να υπάρχει ο σωστό εξοπλισμό, οι σωστέ ικανότητε, Αλλά αυτό δεν αρκεί. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει και πολιτική βούληση. Πολιτική βούληση να χρησιμοποιηθούν τα μέσα αυτά για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις ε, της ασφάλειας που απειλούν την Ευρώπη για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε κρίσεις πιο μακριά από το σπίτι μας, οι οποίες ενδεχομένω να μας επηρεάσουν όμως και για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα το φόρτο αυτό με τους εταίρους μας από τη Βόρεια Αμερική. Προκειμένου λοιπόν να συμβούν αυτά, τα έθνη της Ευρώπης θα πρέπει να αναπτύξουν μια πραγματικά παγκόσμια προοπτική και προσέγγιση. Δεν θα πρέπει να χανόμαστε στα του οίκου μα, στα θέματα που αφορούν μόνο την Ευρώπη. Θα πρέπει το βλέμμα μας να στραφεί προς τα έξω. Και θα πρέπει η Ευρώπη και η Βόρεια Αμερική να συνομιλούν πιο τακτικά, με πιο ανοιχτό και ελεύθερο χαρακτήρα και με μεγαλύτερη ειλικρίνεια. Στο μοναδικό διατλαντικό φόρουμ που ονομάζεται ΝΑΤΟ και μεταξύ ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κλείνοντας λοιπόν, πρέπει να πω ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου θα πρέπει να καταδείξει μια Ευρώπη η οποία είναι και ικανή να δράσει και πρόθυμη να δράσει. Και θα πρέπει να ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ να ενεργούν πιο πολύ από κοινού, να συντονίζονται πιο πολύ, να συζητούν πιο πολύ και να συνεργάζονται πιο πολύ. Προκειμένου να το πετύχουμε αυτό, θα χρειαστούμε έντονη πολιτική αποφασιστικότητα και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Είμαι αισιόδοξο και βέβαιος ότι μπορούμε να έρθουμε στο ύψος των περιστάσεων. Το χρωστούμε άλλωστε στους φορολογούμενους στο εκλογικό μας κοινό. Να τους δώσουμε την καλύτερη δυνατή ασφάλεια Και μετά την εισαγωγή αυτή προσβλέπω σε μια πολύ έντονη συζήτηση σήμερα το απόγευμα. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. Σας ευχαριστούμε κύριε Γενική Γραμματέα και για την ομιλία σας και για την παρουσία σας και χαρήκαμε ιδιαίτερα που είχατε την ευκαιρία να έρθετε για να έχουμε αυτή τη συζήτηση. Ο κύριος Αλαφράγκο πρώτος που ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Φας. Μερικές φορές να καθυστερώ και μετά παραβιάζομαι. Πρώτα κύριος Δανουζάμ. Ευχαριστώ. Χωάνι Γνάσιο. Μην ανησυχείς. Δεν θα θέσω εγώ την ερώτησή σου. Δεν θα σε προλάβω. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Γενικό Γραμματέα για την τακτική, πολύ χρήσιμη και ευπρόσδεκτη πάντα παρουσία του. Και σας ευχαριστώ και για το μήνυμά σας που ήταν απερίφραστο και σαφέστατο σε ό,τι αφορά τις ε, ικανότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και την ε, κοινή στρατηγική ασφάλειας και άμυνας και τη στρατηγική που θέλετε να αναπτυχθεί, μάλιστα με πυγμή. Η ομιλία σας άλλωστε απηχεί την ομιλία που ακούσαμε πριν από δύο χρόνια τον ε, Αμερικανό Υπουργό ε, Άμυνας όταν ήρθε στις Βρυξέλλες που κάλεσε τους ε, Ευρωπαίους να δράσουν περισσότερο και καλύτερα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό και τις ικανότητες. Και είναι και σημαντική δική μας σοβαρή ανησυχία. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, γιατί όλοι γνωρίζουμε τις θεσμικές δυσχέρειες, τις θεσμικές δυσκολίες που υπάρχουν στη σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Γνωρίζουμε επίσης ότι αυτές οι θεσμικές και πολιτικές δυσκολίες δεν πρόκειται να επιληθούν εύκολα και πρόθεσμα. Οπότε, πώς πιστεύετε ότι μπορεί να βελτιωθεί ο συντονισμός μεταξύ των δύο μέρων και κατά τη γνώμη σας, σε τι, ποιο είναι το εξωτερικό πεδίο, ε, το υπάρχον ή το μελλοντικό, ε, πεδία στα οποία μπορούμε να συσφίξουμε τη συνεργασία μας. Μερικοί από εμά, ο Άντριου Ντάφ που είναι εδώ σήμερα, πήγαμε στο Northwood την προηγούμενη εβδομάδα και ε, επισκεφθήκαμε το Γενικό Επιτελείο της Επιχείρησης Ατελάνδης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα ε, συναντήσαμε και τον ε, επικεφαλής ε, του Ναυτικού Επιτελείου του ΝΑΤΟ και διαπιστώσαμε ότι το ΝΑΤΟ έχει πολύ μεγάλες φιλοδοξίες στον Ειδικό ωκεανό. Τι θα γίνει στην περίοδο μετά το Αφγανιστάν, μετά το 2014 λοιπόν και αυτή την επιθυμία τη βούληση του ΝΑΤΟ να βρει πάση θυσία θα έλεγα νέους ορίζοντες. Είναι κάτι λογικό κάτι τέτοιο, συνετό ε, και μάλιστα ε, σωστά διαρθρωμένο σε σχέση με τους υπόλοιπους διεθνείς οργανισμούς. Υπάρχει συνένεση για το θέμα αυτό στο ΝΑΤΟ και σε ποιες ζώνες σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί περισσότερο το ΝΑΤΟ στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Σαλαφράγκα. Θα ήθελα και εγώ να ε, καλωσορίσω τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ στη συνεδρίασή μας. Να του πω καταρχήν ότι Λυπούμαστε ιδιαίτερα για το θάνατο το περασμένο Σάββατο πολλών στρατιωτών της αποστολής του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν και θα ήθελα να σας ε, διαβεβαιώσω ότι συμμεριζόμαστε πλήρως στην ανάλυση σας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι περισσότερο πολιτική και οικονομική παρά στρατιωτική ένωση. Οπότε ή η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αντιμετωπίσει με αποτελεσματικό και αξιόπιστο τρόπο τις διάφορες απειλές ή αλλιώς δεν θα μπορέσει να αναλάβει ή να ανταποκριθεί στις φιλοδοξίες της για παγκόσμιο ηγετικό ρόλο. Έχουμε 1.800.000 στρατιώτες, 500.000 περισσότερες από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρ' όλα αυτά έχουμε προβλήματα και δυσκολίες στο να κινητοποιησουμε 4000 4-5.000 στρατιώτες σε διάφορες επιχειρήσεις της κοινή εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. <clears throat> Έχω δύο ερωτήσεις. Ε, ως προς την πρώτη, θα ήθελα να μου πείτε πώς ε, το ΝΑΤΟ ε, σχολιάζει τη νέα επέμβαση του Ισραήλ στην ε, εμπλοκή στη Συρία και πώς μπορεί να επηρεάσει κάτι τέτοιο ένα μέλος του ΝΑΤΟ που είναι η Τουρκία. Τι διδάγματα μπορούμε να αντλήσουμε από την ζώνη αποκλεισμού πτήσεων της, που εφαρμόσαμε στη Λιβύη μετά τις εξελίξεις ειδικά στη Συρία πιστεύετε ότι μπορεί να εφαρμοστεί αποκλεισμό πτήσεων και στη Συρία δεδομένης της κατάστασης και των συνθηκών που επικρατούν εκεί. Δεύτερον, Συνεχίζοντα την ερώτηση του φίλου και συναδέλφου κ. Ντανζάν, θα ήθελα να ρωτήσω τι, γίνεται, τι θα γίνει στο Αφγανιστάν μετά το 2014 και ποιο θα είναι ο ρόλο που θα δώσουν οι αρχέ τη χώρα στο ΝΑΤΟ στην Ατλαντική Συμμαχία. Επίσης, ε, θα ήθελα να σας ρωτήσω με ποιο τρόπο ε, εργάζεται και πώς προσπαθεί το ΝΑΤΟ να συνδυάσει αυτό το Smart Defense, την έξυπνη άμυνα, με την πολιτική του pooling and sharing που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο συνάδελφος κύριος Κλίχτ ε, με τριπλή ιδιότητα. Είναι πρώην μέλος ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μέλος της ε, Γερουσίας Πολωνίας και πρώην Υπουργός Άμυνας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να σας πω ότι είναι μεγάλη χαρά για μένα το ότι μπορώ να ξαναβρίσκομαι εδώ και το ότι μπορώ να μιλήσω για τη συμβολή της Ευρώπης στο ΝΑΤΟ και στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω τρεις παρατηρήσεις. Πρώτον, όσον αφορά στη συνέχιση της ε, δραστηριότητας του ΝΑΤΟ, όχι μόνο σε επιχειρήσεις, αλλά και σε θέματα ασφάλειας ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί η στρατηγική αυτή ενδέχεται να οδηγήσει στο να υπάρξει αποδυνάμωση της ασφάλειας στην Ευρώπη. Θεωρώ λοιπόν είναι σαφές ότι στην Ευρώπη. Η Ευρώπη καλείται να προσφέρει περισσότερα στο θέμα του ε, δυναμικού και των επιχειρήσεων. Οι Αμερικανοί μετά την αλλαγή των προτεραιοτήτων και τη στρατηγική που εξέφρασαν στις αρχές ε, του προηγούμενου έτους. Όπως επίσης ε, και το γεγονός ότι μετέθεσαν πλέον στις προτεραιότητές τους από τη Μέση Ανατολή προς τον Ειρηνικό, οι Αμερικανοί περιμένουν μεγαλύτερη συμβολή της Ευρώπης. Και η δική μου ερώτηση είναι η εξής. Αυτή τη στιγμή πώς ακριβώς αξιολογείται την ε, έξυπνη άμυνα. Είναι μια πρωτοβουλία καθοριστικής σημασίας που ανελήφθη πέρυσι κατά τη διάρκεια της ε, συνάντησης κορυφής και αποτελεί μια απάντηση για την κρίση που αποτελούν οι δυνατότητές μας. Τώρα όσον αφορά τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ υπάρχει ένας μόνιμος διάλογος μεταξύ ημών και της κυρίας Αστόν ε, θεσμοθετήθηκε πριν από κάποια χρόνια πρόκειται για ένα διάλογο εργασίας ε, χωρίς να ε, έχει θεσμοθετηθεί θεωρώ όμως ότι πρέπει να διατηρηθεί προς όφελος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του ΝΑΤΟ και ρωτώ λοιπόν ε, κατά την άποψή σας, πώς πρόκειται να εξελιχθεί ο διάλογος αυτός. Η τρίτη μου παρατήρηση αφορά την αναγκαιότητα συνεργασία ε, ανάμεσα στους φορείς ACT και την Υπηρεσία Εξωτερικής ε, Δράσης. Αυτό είναι απαραίτητο και όσον αφορά στις δυνατότητες ορισμένων κρατών μελών. Κυρίως στον τομέα του περίφημου pooling and sharing και της έξυπνης άμυνας. Μέχρι ποιο βαθμό λοιπόν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι οι δύο αυτές ε, πρωτοβουλίες ε, έχουν εναρμονιστεί γιατί θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει αυτή η εναρμόνιση. Κυρία Γιακονσάρη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήταν ε, πολύ ενδιαφέρουσα η ομιλία σας κύριε Γενική Γραμματεύ. Μας είπατε ότι το ΝΑΤΟ είναι ένα μοναδικό φόρουμ διατλαντικό, διατλαντικού διαλόγου και είναι αναφυσβήτητο κάτι τέτοιο, σε αυτός ο χαρακτήρας του ΝΑΤΟ και θεωρώ ότι είναι πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι το ΝΑΤΟ επικεντρώθηκε στις ε, νέες ασφάλειες ε, όπως είναι οι ασφάλεια στον κυβερνοχώρο επικρατεί η γνώμη ότι το ΝΑΤΟ είναι μερικές φορές κάτι το καινούριο της μόδας, ε, γιατί αρχίζει, αρχίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και γίνονται πιο εσωστρεφείς ε, και αυτό κάπως υποβάθμισε το ΝΑΤΟ. Ερωτώ λοιπόν σας, πιστεύετε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αρχίζουν και αδιαφορούν ή χάνουν κάπως το ενδιαφέρον τους για την Ευρώπη. Και η δεύτερη μου ερώτηση αφορά το pooling and sharing και τον ευρωπαϊκό ενθουσιασμό που επικρατεί για αυτό το θέμα της κοινή διαχείρισης των πόρων. Και στο ΝΑΤΟ και σε κάποια ερευνητικά Ινστιτούτα που πρόσκειται στο ΝΑΤΟ γίνονται έρευνες για το πόσα χρήματα των φορολογουμένων χρησιμοποιούνται για να συντηρηθούν κάποια παλιά κτίρια, παροχημένος εξοπλισμός και κάποιες ε, δομές άμυνας που είναι και αυτές απειρχιωμένες. Εν μέσω μάλιστα της ε, οικονομικής κρίσης θεωρώ ότι θα πρέπει να δείξουμε περισσότερο ενθουσιασμό για την κοινή διαχείριση των πόρων, για αυτό το pooling and sharing. Έγινε κάποια έρευνα σχετικά για να αποτιμηθούν τα κονδύλια τα δημόσια κονδύλια που σπαταλούνται με τον τρόπο αυτό για τη συντήρηση παροχημένων κτηρίων ή εξοπλισμών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ για... Τι γίνεται, δεν λειτουργεί το μικρόφωνο μου. Α, μάλιστα, βρήκα άλλο. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ για την ε, συνοπτική αλλά μεστή και πολύ σημαντική παρέμβασή του που μίλησε για την ανάγκη να επενδύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ περισσότερο στην ασφάλειά της. Και μάλιστα όντως ε, στα πλαίσια του ΝΑΤΟ το θέμα του burden sharing, της κατανομής ε, του βάρους ε, είναι, δεν είναι κάτι καινοφανές. Μάλιστα προηγείται ακόμη και τις πτώσεις του τείχους του Βερολίνου το θέμα αυτό. Έχουν περάσει όμως τόσα χρόνια και διαπιστώνουμε ότι δυστυχώς ε, δεν έγιναν κάποιες ε, ρηξικέλευθες αλλαγές. Βρισκόμαστε σήμερα σε μια κατάσταση όπου βλέπουμε τις είπα να μεταθέτουν το επίκεντρο του ενδιαφέροντός τους προς τον ειρηνικό. Μάλιστα επέστρεψα άρτη από μια αποστολή στην Ινδία που αν θέλω να πω με μια φράση ε, ποια είναι η, η αίσθηση του πολιτικού κόσμου των Ινδιών για την Ευρώπη είναι ότι η Ινδία πιστεύει, έχει πίστη στις μεγάλες χώρες, έχει πίστη στι Ηνωμένε Πολιτείε. δεν έχει καμία πίστη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα λέω κάποιου συνοπτικά και χονδροκομμένα, αλλά σε γενικέ γραμμέ αυτό είναι το μήνυμα που λάβαμε στην Ινδία. Τώρα, οι απειλέ που μα περιστοιχίζουν είναι πιο σημαντικέ και σοβαρέ από ποτέ, παρόλο που μερικέ φορέ δεν το αντιλαμβάνεται αυτό η κοινή γνώμη. Και η κατάσταση στη Συρία, όπου φυσικά μια στρατιωτική επέμβαση είναι απευκταία, αλλά πολύ υπάρχει μεγάλο κίνδυνο να γίνει απαραίτητη μια τέτοια στρατηγική επέμβαση, αν κάποιο βάλει χέρι στα χημικά όπλα. Και από αυτή την άποψη θα, ήθελα, θα θέλαμε να ακούσουμε κάποια πιο αποφασιστικά σχόλια, να δούμε μεγαλύτερη αποφασιστικότητα. Και στη διάσκεψη κορυφή που θα αφιερωθεί στην ε, ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ΝΑΤΟ θα απευθύνει έκκληση προς την Ευρώπη ως ΝΑΤΟ ε, να δημιουργηθεί μια πραγματική ευρωπαϊκή άμυνα. Γιατί τη στιγμή που περικόπτονται οι κρατικοί προπολογισμοί και τα αμυντικά μέσα και που η Γαλλία και, οι Ηνωμένες, ε, και το Ηνωμένο Βασίλειο κάνουν κάποιες καταστροφικές επιλογές στρατιωτικές, αν αφήσουμε τον καθένα να λειτουργήσει με βάση την εθνική του σημαία, δεν θα απομείνει τίποτα αξιόπιστο πια στην άμυνα στην Ευρώπη. Νομίζω ότι είναι η στιγμή να συνενώσουμε τα μέσα μας, πολλό δε μάλλον που περικόπτονται οι προπολογισμοί μας. Και παρόλα αυτά, στα εθνικά κοινοβούλια δεν ακούμε ε, τέτοια επιχειρηματολογία στα πλαίσια της οικονομικής ε, κρίσης που βιώνουμε. Παρόλα αυτά είναι απολύτως απαραίτητο κάτι τέτοιο. Οπότε το ΝΑΤΟ θα θέσει με ζαφήνει αυτό το θέμα, αυτή την έκκληση, θα κάνει αυτή την έκκληση, θα, θέσει, θα λάβει αυτή τη θέση με αποφασιστικότητα. Γιατί Φυσικά θέλουμε, ε, και εγώ ήμουν ανέκαθεν υπέρ του να έχουμε περισσότερε δράσει στα πλαίσια του ΝΑΤΟ ω χώρε. Μήπω το ΝΑΤΟ όμω θα ζητήσει ενσωμάτωση των στρατιωτικών μέσων ε, των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε. Ευχαριστώ κύριε Σντάφ. Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Δύο σημεία ήθελα να δείξω. Καταρχάς, καταλαβαίνουμε ότι ένα μεγάλο εμπόδιο στις συνεργασίες μεταξύ ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι πάντα το Κυπριακό. Συμφωνείτε μαζί μου ότι γι' αυτό θα ήταν σωστό και ενδεικνυόμενο να ζητηθεί από τον Τούρκο Πρωθυπουργό Ρετζεπταυγή Περντογάν να παρευρεθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου. Νομίζω ότι αν του ζητηθεί να παρευρεθεί θα έχει την πρώτη του ευκαιρία να μιλήσει σε ομότιμους από το 2004. Και έχει περάσει πολύ καιρό από το 2004. Κατά δεύτερον, μετά από μια επίσκεψη στο Northwood που ανέφερε και ο κύριος Νταντζάν. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια για την προσέγγιση του ΝΑΤΟ σε ό,τι αφορά το μέλλον του προγράμματος Αταλάντη. Σε ό,τι αφορά το θέμα της πειρατείας στη Σομαλία. αν ε, σταματήσει μέχρι τα τέλη του επόμενου έτους η επιχείρηση, οι πειρατές θα επιστρέψουν. Και πιστεύετε ότι θα μπορούσαμε να διδαχτούμε από αυτά που έχουν γίνει και από την επιτυχία που σημειώθηκε στην επιχείρηση της Σομαλίας. σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη παρά, παρόμοιων ναυτικών δυνάμεων. Στον κόλπο της Γουινέας. Ευχαριστώ. Thank you very much indeed. Σας ευχαριστώ Relevant, um, uh, για τις πολλές και εύστοχες ερωτήσεις. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω κύριε Ντανζόν για τα ευγενικά σας λόγια. Με ρωτήσατε πώς θα μπορούσαμε να συντονίσουμε με καλύτερο τρόπο τις δράσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Και ο κύριος Κλίχ έθεσε σχετικά ερωτήματα. Νομίζω ότι τρει είναι οι τομείς στους οποίους θα πρέπει να υπάρξει πολύ στενή συνεργασία και πολύ στενό συντονισμό μεταξύ ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, Καταρχά σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις. Από κοινού διοργανώνται οι επιχειρήσει στο Αφγανιστάν, στο Κωσυφοπαίδιο και θα πρέπει να σας πω ότι παρά τα πολιτικά προβλήματα που υπάρχουν, ε, εν πάση περιπτώσει, ας τα πούμε προβλήματα, να τα πούμε προκλήσεις σε ό,τι αφορά το συντονισμό μας και στη συνεργασία μας, καταφέρνουμε να συντονιστούμε ομαλά Επιτόπου Η EUPOL και η ISAF συνεργάζονται αποτελεσματικά. Στο Αφγανιστάν η KFOR και η ULEX συνεργάζονται πολύ αποτελεσματικά στο κοσίφο πεδίο και συνδράμουν η μία τη άλλη την άλλη. Άρα θεωρώ ότι καθημερινά στι καθημερινέ μα επιχειρήσει καταφέρνουμε να συνεργαστούμε. Κατά δεύτερον, χρειάζεται στενό συντονισμό σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη των ικανοτήτων μα, των δυνάμεών μα. Και αυτό με οδηγεί στι ερωτήσει σε ό,τι αφορά την έξυπνη άμυνα, το pooling and sharing, το οποίο αναφέρθηκε από διαφόρου. Ο κ. Σαλαφράγκα μίλησε για το pooling and sharing και για την ευφυή άμυνη και ο κ. Κλίχ αναφέρθηκε σε αυτά. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν δημιουργούνται παράλληλα προγράμματα. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα προγράμματα είναι συμπληρωματικά και ότι ε, αξιοποιούν με τον σωστό τρόπο τα χρήματα των φορολογουμένων. Να μην υπάρχει ε, αλληλεπικάλυψη, να μην υπάρχει ανταγωνισμός ε, μη παραγωγικός. Και θα μπορούσα να σας δώσω ένα εξαιρετικό παράδειγμα για το πώς κάναμε μια παραγωγική κατανομή του φορτίου. Στο, στην σύνοδο στο Σικάγο του προηγούμενου έτος, οι ευρωπαϊκοί σύμμαχοι δεσμεύτηκαν να αναπτύξουν ικανότητες σε ό,τι αφορά ανεφοδιασμό στον αέρα, παρόλο ότι υπάρχει σχετική ικανότητα στο ΝΑΤΟ σε ό,τι αφορά τον αέριο ανεφοδιασμό. Εξαρτόμαστε όμως από τις, ε, τον εξοπλισμό των Αμερικανών. Χρειαζόμαστε λοιπόν και σχετικό ευρωπαϊκό εξοπλισμό. Έγινε λοιπόν αυτή η δέσμευση από τους Ευρωπαίους Συμμάχους στο Σικάγο και αυτό αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα για το πώς μπορεί να υπάρχει κατανομή ε, του φορτίου. Δεν υπάρχει λόγος να το κάνει αυτό το ΝΑΤΟ. Και κατά τρίτον χρειαζόμαστε πιο πολύ συνεργασία και διαβούλευση και συντονισμό σε ό,τι αφορά την πολιτική. Και εδώ πραγματικά η κατάσταση είναι παράλογη στις επίσημες συναντήσεις μπορούμε και μας επιτρέπεται να συζητάμε μόνο ένα θέμα. Ένα θέμα. Γιατί τη Βοσνία. Γιατί υπάρχει το σχετικό πλαίσιο που το ορίζει αυτό. Δεν θα επισέλθω σε τεχνικές λεπτομέρειες. Το αποτέλεσμα είναι ότι μόνο αυτό το θέμα μας επιτρέπεται να συζητάμε στις επίσημες συναντήσεις. Και οι συναντήσεις αυτές Λαμβάνω χώρα με την Ευρωπαϊκή Ένωση με τα 26 μέλη, χωρίς τη συμμετοχή των Κυπρίων. Και για τον ίδιο λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλει να διοργανώνει πολλές συναντήσεις με 26 μόνο από τα 27 κράτη-μέλη. Και αν ε, δεχόμασταν να συζητήσουμε άλλα θέματα τα οποία είναι σχετικά, όπως το 25 για παράδειγμα, αυτό μπορεί να γίνεται μόνο σε άτυπες συναντήσεις και στις περιπτώσεις αυτές ε, ε, αντιδρούν οι Τουρκοί και δεν δέχονται να υπάρχουν πολλές τέτοιες συναντήσεις. Εκεί βρισκόμαστε και άρα εάν δεν βρούμε μία λύση για το Κυπριακό, εάν δεν βρούμε μία λύση για το Κυπριακό, θα συνεχίσει αυτό το θέατρο του παραλόγου. Εδώ λοιπόν είναι ένα θέμα στο οποίο θα πρέπει να κινηθούμε προς το ευρώ, να σημειώσουμε πρόοδο. Έχω προτείνει στο παρελθόν κάποιες ε, προτάσεις, κάποιες λύσεις, αλλά διαπιστώνω ότι η τελική πολιτική λύση προαπαιτεί μία προσέγγιση των μερών στην Κύπρο και θα έπρεπε να γίνει αυτό γιατί είναι τεράστιες οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Έχουν φυσικούς πόρους τους οποίους θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν μετά την επανένωση της νήσου. Και εδώ θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να δραματίσει σημαντικό ρόλο. Θεωρώ ότι έχει κάποια αμόχλευση η Ευρωπαϊκή Ένωση για να διευκολύνει την εξέφραση μια λύση στο πρόβλημα αυτό. Ο κ. Ντανζάν επίσης με ε, ρώτησε τι θα γίνει με τον άτομο μετά το 2014. Κατά πόσον ε, αναζητούμε νέα καθήκοντα, κατά πόσον θέλουμε να εφεύρουμε νέες ε, δραστηριότητες και ενέργειες προκειμένου να συνεχίσει να έχει σημασία το ΝΑΤΟ. Σε καμία περίπτωση δεν συμβαίνει αυτό. Δεν χρειάζεται σε καμία περίπτωση να εφεύρουμε το οτιδήποτε. Είμαστε υπεραπασχολημένοι με αυτά που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Άρα το ΝΑΤΟ μετά το 2014 θα είναι ένα ΝΑΤΟ το οποίο θα είναι σε θέση και θα είναι προετοιμασμένο να δράσει αν χρειαστεί. Και ένας τρόπος να γίνει αυτό θα είναι διασφαλίζοντας ότι η ικανότητα που έχουμε αναπτύξει για συνεργασία στο Αφγανιστάν, αυτή η ικανότητα λοιπόν θα αναπτυχθεί περισσότερο στο μέλλον. Πρωτοβουλία Connected Forces το ονομάζουμε σε ό,τι αφορά όλες τις ασκήσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αυτά που μάθαμε λοιπόν στο Αφγανιστάν θα συνεχίσουν να υπάρχουν ακόμα και όταν αποσυρθούμε από το Αφγανιστάν. Και πιστέψτε με θα ανακύψουν και να θα αναντηθούν νέες ε, υποχρεώσεις, νέα καθήκοντα και εμείς είμαστε έτοιμοι για το αναπάντεχο. Αν ε, με ρωτούσατε όταν ανάλαβε τα καθήκοντά μου το, Αύγουστο του 2009, αν μπορούσα να φανταστώ το ΝΑΤΟ στην Λιβύη, σίγουρα θα σας απαντούσα αρνητικά. Παρ' αυτά όμως, ανέκυψε ως καθήκον, ε, καθήκον στο οποίο κληθήκαμε να ανταποκριθούμε και αυτό ακριβώς ε, τονίζω ότι θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το αναπάνταχο. Και αυτό θα είναι το καθήκον μας για μετά το 2014. Για τον κύριο Σαλαφράγκα το ίδιο ρωτήσατε ακριβώς. Επίσης, ο κ. Σαλαφράγκα μου έθεσε μία ερώτηση για τη Συρία. Και για την Ισραηλινή επίθεση στη Συρία. Είδα το σχετικό ανακοινωθέν τύπου. Δεν έλαβε χώρα οποιαδήποτε τέτοια δραστηριότητα σε περιοχές σχετικές σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη πυράβλων ε, πάτριο στην Τουρκία. Αλλά προφανώς μας απασχολεί η καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση μας ε, ε, απασχολεί το ενδεχόμενο ε, διάχυσης του κινδύνου στην περιοχή μας, απασχολεί το ενδεχόμενο χρήσης ε, πυρηνικών χημικών όπλων. Άρα καλούμε την διεθνή κοινότητα να βρει μια λύση το συντομότερο δυνατόν. Και αυτό θα σήμαινε ότι θα πρέπει να βρεθεί συμφωνία μεταξύ των πέντε μόνιμων μελών του, Ευρωπαϊκού, του ε, Συμβουλίου Ασφαλείας του ΝΑΤΟ. Ο μοναδικό τρόπο να επιληθεί το θέμα είναι με πολιτική βούληση, αλλά χρειαζόμαστε ε, ισχυρά και δεσμευτικά μέτρα από την διεθνή κοινότητα. Ο κύριος Κλίχ με ρώτησε κατά πόσον τη μετάθεση της, των ΗΠΑ στην Αυστρία ε, θα είναι καθοριστική. Αυτό θα εξαρτηθεί από εμάς τους Ευρωπαίους, απαντώ. Είναι προς το συμφέρον μας ε, οι ΗΠΑ να ξαναζυγίσουν και να εξισορροπήσουν τα συμφέροντά τους και σε ό,τι αφορά και τα δικά μας συμφέροντα στην ε, Νοτιοανατολική Ασία. Αλλά αν θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι Αμερικανοί θεωρούν ισότιμο εταίρο την Ευρώπη, η Ευρώπη θα πρέπει να επενδύσουν και αυτοί με τη σειρά τους στην διατρατική αυτή σχέση πολιτικά, οικονομικά αλλά και στρατιωτικά. Η κυρία Γεκονσάρη έθεσε ουσιαστικά το ίδιο ερώτημα. Κατά πόσο ο ρόλος των ΗΠΑ στην Ασία θα υπονομεύσει τον ΝΑΤΟ. Όχι καθεαυτός. Αλλά ασφαλώς αν οι Ευρώπη δεν επενδύσουν στην ιδρυτική σχέση, ενδεχομένως να τους αποδυναμώσει, να μας αποδυναμώσει. Αλλά είδαμε ότι είναι ισχυρή η δέσμευση των ΗΠΑ στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. Για παράδειγμα, η συμβολή την ΗΠΑ για ένα ευρωπαϊκό αντιπραυλικό σύστημα πρόκειται για μία δέσμευση των ΗΠΑ για να ανταποκριθούν σε ανερχόμενες, αναδυόμενες μελλοντικέ προκλήσεις. Αντί να υπάρχουν λοιπόν πολλές ε, μόνιμα σταθμευμένες ε, δυνάμεις στην Ευρώπη, οι ΙΠΑ τώρα αναζητούν σύγχρονους τρόπους για να ανταποκριθούν στις ε, προκλήσεις του σήμερα. Και αυτή την άποψη ε, με ρωτήσετε τι γίνεται με τις ε, παροχημένες δομές, τις, τον απειρχιωμένο εξοπλισμό, τα κτίρια κτλ. Αν έχουμε έρευνες για το πόσα χρήματα ξοδεύονται σε τέτοιες ε, απειρχιωμένες, ε, πεπαλαιωμένες δομές. Δεν γνωρίζω να έχει γίνει τέτοια έρευνα. Αλλά πραγματικά θέλουμε να μεταρρυθμίσουμε τις στρατιωτικές μας δυνάμεις προκειμένου να έχουμε ευκολότερη ανάπτυξη, λιγότερο στατικές ε, δομές και πιο κινητικές, πιο ευέλικτες για να γίνεται ανάπτυξή τους όπου κρίνεται απαραίτητο. Και αυτή είναι η υπεπτουσία των συνεχιζόμενων προσπάθειών μας ε, για μεταρρύθμιση και μεταμόρφωση του ΝΑΤΟ. Ο κύριος Τέικερ ε, με ρώτησε ευθέως αν το ΝΑΤΟ θα συστήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει μια ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας. Ως Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ δεν πρόκειται να επέμβω εγώ στις ε, ενωσιακές πολιτικές. Πιστεύω πάντως και ακούσατε τη σημερινή μου ομιλία. Πιστεύω λοιπόν ότι θέλουμε μια πιο ενισχυμένη ευρωπαϊκή άμυνα και δεν βλέπω καμία αντίφαση μεταξύ ενό ισχυρού ΝΑΤΟ και μια ισχυρή αμυντική συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίθετα, πιστεύω ότι έτσι θα ενισχυθεί ο κοινοτικό πυλώνα εντό του ΝΑΤΟ. Οπότε, αν έχουμε μια ενισχυμένη αμυντική πολιτική στην Ευρώπη, σημαίνει ότι θα επιδίσουμε περισσότερο στι στρατικέ μα ικανότητε. Και το λέω και εγώ ευθέω και ανοιχτά. Και όχι σε νέε γραφειοκρατικέ δομέ και σε, σε νέου θεσμού. Τότε πραγματικά θα έχουμε μια χρήσιμη συμμετοχή και συμβολή στην ενίσχυση της παγκόσμιας ασφάλειας. Αλλιώς θα είναι έπεπτερόεντα και μια τρύπα μες στο νερό, όπως είπα και πριν. Είπε υπέρ, αλλά δεν πρόκειται να επέβω λοιπόν, συνοψίζοντας. Επίσης, για να ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό, πολύ συχνά συζητούμε και ξέρω ότι και οι πολιτικές ομάδες ε, εξετάζουν το κατά πόσο χρειαζόμαστε μια κοινή ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική. Νομίζω ότι από ρεαλιστική άποψη δεν πιστεύω θα το ζήσουμε αυτό, θα το δούμε με τα μάτια μας εμείς, ότι θα είμαστε ζωντανοί για να δούμε κάτι τέτοιο. Και παρόλο που θεωρώ ότι είμαι σχετικά μακρόβιος, θα ζήσω αρκετά χρόνια ακόμη. Πάντως, ως Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ έμαθα πόσο ε, τα έθνη κράτη προασπίζουν την ακαιρεότητά τους και την εθνική τους κυριαρχία σε ό,τι αφορά τα αμυντικά θέματα και τα θέματα ασφάλειας. Είναι σχεδόν θέμα ταμπού για τα κράτη αυτό το θέμα. Και το προασπίζουν πάση θυσία ως αποκλειστική αρμοδιότητα. Δεν πιστεύω λοιπόν ότι θα υλοποιηθεί κάτι τέτοιο στο εγγύς μέλλον. Πάντως πιστεύω ότι ε, τα κράτη παρόλα αυτά θα ενισχύσουν τη διασυνοριακή του συνεργασία γιατί τους χρειάζεται κάτι τέτοιο. Οπότε θα δούμε όλο και περισσότερα πολυμερή σχέδια και σχέδια. Όπως και να τα πούμε, ε, smart defense, έξυπνη άμυνα, pooling and sharing, συνένωση και κοινή διαχείριση των πόρων, σίγουρα θα υπάρχουν. Αλλά δεν θα μπορέσει η χώρα να αγοράζει πανάκριβους αμυντικούς εξοπλισμούς. Ακόμη και οι πλούσιες χώρες ε, θα χρειαστεί να συνεργαστούν. Και από αυτή την άποψη θα έχουμε όλο και περισσότερες ε, συλλογικές αμυντικές προσπάθειες στην Ευρώπη τα επόμενα χρόνια. Άντριου Νταφ, με ρωτήσατε κατά πόσο θα ήταν καλή ιδέα να προσκαλέσουμε τον Πρωθυπουργό Ερτογάν στο Συμβούλιο Κορυφής του Δεκεμβρίου. Δεν πρόκειται εγώ να επέμβω στις ευρωπαϊκές αποφάσεις για το ποιο θέλουν να προσκαλέσουν στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια. Και τέλος, για την πειρατεία, ήταν όντως επιτυχημένη αυτή η επιχείρηση και το μάθημα που διδαχθήκαμε είναι ότι μια στενο, ένα στενός διεθνής συντονισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΝΑΤΟ και μεμονωμένων φορέων μας επιτρέπει να επιδείχουμε πάρα πολλά πράγματα. Και δεν αποκλείεται, με βάση αυτά τα διδάγματα που αντιλήσαμε, να κρίνουμε ότι μπορούμε να αναπτύξουμε ε, σκάφη μας ε, πολεμικά πλοία και σε άλλες περιοχές του κόσμου, σε μια διεθνή προσπάθεια για να εξασφαλίσουμε ε, ελεύθερος από πειρατεία θαλάσσιας διόδους. Γιατί η πειρατεία δεν θα περιοριστεί μόνο στη Σομαλία, πολύ πιθανόν να ανακύψει και σε άλλες θάλασσες. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω το λόγο σε κάποιον που επιθυμεί να σχολιάσει τις παρατηρήσεις που κάνατε σχετικά ε, με τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-ΝΑΤΟ ε, και το ότι είναι απαραίτητο να υπάρχουν οι σχέσεις αυτές ε, Κύριε παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαστε σήμερα εδώ κύριε Γενική Γραμματέα. Είναι πολύ ευχάριστο το να έχει κανείς ε, και κάποιο τόνο πραγματικότητας ε, ρεαλισμού σε αυτό το θεσμό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είπατε ότι το ΝΑΤΟ μετά το 2014 δεν χρειάζεται να επανακαλύψει τον τροχό, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση καλύτερα να το ε, πράξει αυτό πράττει αυτό συνεχώς, ε, προσπαθεί να αναζητήσει ευκαιρίες ε, έτσι ώστε να ε, δικαιολογήσει την ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας. Έχω λοιπόν την εντύπωση ότι το ερώτημα που πρέπει να τεθεί είναι το εξής. Πώς πρέπει να ενισχυθούν οι δυνατότητες των δημοκρατιών, οι δυνατότητες τους να δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον επικίνδυνο κόσμο και όχι το πώς μπορούμε να αιτιολογήσουμε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ξέρετε κύριε Γενική Γραμματέα, καταλαβαίνω ότι είστε σε πολύ δύσκολη θέση. Είσαστε ένα είδος διπλωμάτη που παρεμβαίνει και στην πολιτική. Ε, κατ' ουσίαν όμως είστε διπλωμάτης. Δηλαδή ε, καλείστε να μιλήσετε με ένα τέτοιο τρόπο ώστε κανένα από τα 28 κράτη-μέλη σας να μην προσβληθεί. Παραμένει βέβαια το γεγονός ότι ε, εδώ μιλάμε για κάτι διαφορετικό. Δεν μιλάμε για την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων, αλλά το να αναζητηθεί ένας ε, ρόλος ε, για να μπορεί να δράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πιστεύετε τώρα που δεν υπάρχουν αρκετοί πόροι αντί η Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργεί παράλληλους ε, θεσμούς και δομές, θα ήταν καλύτερα να εστιάσει κανείς τις ευρωπαϊκές του προσπάθειες μέσα στο ΝΑΤΟ, γιατί τελικά αυτό θα γίνει. Και όλη αυτή η επικάλυψη των προσπαθειών οδηγεί στο κατ' ουσίαν τα ίδια τα κράτη-μέλη ε, μιλούν μεταξύ τους και πάντα στις ίδιες πόλεις. Αυτή τη στιγμή, όσο εξελίσσονται τα πράγματα, εμένα με ανησυχεί το εξή. Δεν υπάρχει ουσιαστική συζήτηση η συζήτηση που γίνεται εδώ είναι για ρόλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως στην πραγματικότητα αυτό που θέλει κανείς να πει είναι σταματήστε να παίζετε με την πολιτική, ή να φτιάχνετε θεσμούς και δομές, δημιουργήστε περισσότερες δυνατότητες. Αυτό χρειαζόμαστε. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί ο στόχος της είναι τελείως διαφορετικός. Εσείς ε, δεν ανησυχείτε με το ενδεχόμενο αποδυνάμωσης της ε, συμμαχίας, δηλαδή θα έχουμε μια διτή δομή από τη μια την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την άλλη τους Βορειοαμερικανούς. Και γνωρίζω ότι υπάρχουν εδώ άνθρωποι υπέρμαχοι του βορειοατλαντισμού σε αυτό όλο το κύκλωμα που το επιθυμούν κάτι τέτοιο, που θεωρούν αυτός είναι ο στόχος τους. Και ε, για μένα τουλάχιστον αυτή είναι μια πολύ επικίνδυνη κατεύθυνση. Με ενδιαφέρει λοιπόν διακαώς η άποψή σας ε, σχετικά με αυτό τον ενδεχόμενο που ανέφερα. Και επίση, κύριε Γενική Γραμματέα, αυτό που θα ήθελα να κάνετε είναι να ενταρρύνετε τις ευρωπαϊκές χώρες να ε, τοποθετήσουν τις δυνάμεις τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να μην έχουμε μια συνεχή επικάλυψη, ε, να μην δημιουργούν συνεχώς νέες δομές, ε, υποτίθεται εκεί που δεν υπάρχουν. Τον κύριο Ράσμουσεν τον έχω ζήσει πολλές φορές ως Δανό ε, πρωθυπουργό και Προεδρεύοντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ξέρετε εγώ ποτέ δεν τον αντιμετώπισα ως διπλωμάτη. Η κυρία Κόμμπερκ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δίνετε για διάλογο με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Θα ήθελα να επικεντρωθώ στη Ρωσία και την αντιπυραυλική ασπίδα. Θα θυμάστε ότι στη Λισαβόνα με την μεγάλη αυτή φιλία Ρωσίας και ΝΑΤΟ και τις δηλώσεις για συνεργασία σε θέματα αντιπυραυλικής άμυνας. Έκτοτε όμως αντιμετωπίσαμε προβλήματα σε αυτά τα θέματα της αντιπυραυλικής άμυνας. Ποιος είναι ο απολογισμό σα. Τώρα που οι Αμερικανοί ακύρωσαν την τέταρτη φάση της αντιπυραυλικής ασπίδας, διανοίγονται νέε δυνατότητες συνεργασίας με τη Ρωσία για τα θέματα αυτά της αντιπυραυλικής άμυνας. Και τι γίνεται στο Συμβούλιο ΝΑΤΟ Ρωσίας. Είμαι η πρόεδρος της ε, για τη σχέση με το Ιράν και είπατε ότι ίσως ε, το ΝΑΤΟ θα πρέπει να διαδραματίσει κάποιο ρόλο στο Ιράν. Υπάρχουν σχετικά σχέδια και ποιος ήταν ο ρόλος του ΝΑΤΟ στην περίπτωση του Ιράν. Ε, καταρχήν ήθελα να, να σημειώσω, ο κύριος Ράσμουσεν συχνά επικαλείται τους φορολογούμενους και το κοινοβούλιο και τους πολίτες κτλ. Ε, έχουμε στην ε, γνώμη και τη θέση ότι αυτό γίνεται κυρίως για λόγους προπαγάνδας και όχι για λόγους ουσίας και αυτό ε, το λέω για τον εξής λόγο. Γίνεται λόγος παραδείγματο χάρη για μείωση εξοπλισμών. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή όλοι ξέρουμε ότι δρομολογούνται, εφαρμόζονται χρησιμοποιούνται νέα οπλικά συστήματα όπως τα μη επανδρομένα αεροπλάνα, τα drones τα λεγόμενα, τα οποία σκοτώνουν κόσμο πάρα πολλού και στο Αφγανιστάν και σε άλλα μέρη. Το ΝΑΤΟ δεν έχει πάρει καμία θέση για το ζήτημα αυτό. Φυσικά το ενισχύει. Δεύτερο ζήτημα, κυρίε Γενική Γραμματέα. Ε, νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε τι εννοείται με την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Βραχίωνα του ΝΑΤΟ. Και απορώ γιατί δεν το λέτε είναι απλά τα πράγματα για όποιον βλέπει τις καταστάσεις. Το ΝΑΤΟ θέλει να έχει το πρώτο λόγο να επιλέγει εκείνο σε ποιες κρίσεις, σε ποιες διενέξεις θα επεμβαίνει και εκεί που δεν θέλει να πηγαίνει το ΝΑΤΟ ας πάνε οι Ευρωπαίοι. Απόδειξη γι' αυτό είναι αυτό που μας είπατε για το αεροπλάνο ενεφοδιασμό στον αέρα. Εάν υπήρχε κοινή διάθεση και κοινή θέση θα υπήρχε συνεργασία. Αλλά δεν θα υπάρχει συνεργασία, κύριε Γενική Γραμματέα, γιατί υπάρχουν πολύ μεγάλα αντικρουόμενα συμφέροντα μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων, μεταξύ των μεγάλων υπεριαλιστικών δυνάμεων και βεβαίως οι Ηνωμένε Πολιτείε θα χρησιμοποιούν το προνόμιο που έχουν με το ΝΑΤΟ και με το ότι οι συνθήκες, κύριε Νόρντεν, είναι, στην Ουάσιγκτον, όπως ξέρετε, και δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα στο ΝΑΤΟ αν δεν αλλάξει η ιδρυτική συνθήκη ε, του ΝΑΤΟ και γι' αυτό το λόγο οι ΗΠΑ θα έχουν πάνω το πάνω χέρι και προφανώς επειδή δυσκολεύουν τα πράγματα όπως γινόταν παλιά στη Γαλλία με μπόμπου λοριό λένε στους Ευρωπαίους τώρα πάτε εσείς στο Μάλι ή πάτε εσείς δεν ξέρω εγώ πού για να έχω εγώ ελεύθερα χέρια σε άλλα μέτωπα. Τρίτο ζήτημα κύριε Γενική. Πάλι επειδή μιλήσατε για χρήματα των φορολογουμένων και των εργαζομένων και των λαών. Ε, δεν νομίζω τώρα, μιλάμε στα σοβαρά, όταν 20 χρόνια μετά τον πόλεμο στη Ιουκοσλαβία συνεχίζεται η κατοχή του Κωσόβου χωρίς να ξέρουμε πότε θα τελειώσει αυτό το παραμύθι με την ατοική κατοχή στο Κόσοβο ή πότε θα τελειώσει η komme zu Ende, mein ich Και πότε θα τελειώσει το παραμύθι στην, ε, στο Αφγανιστάν. Πολύ περισσότερο που διαβάσαν όλοι τι γινόταν με τη CIA, ποιον χρηματοδοτούσε και για ποιο λόγο πρέπει να, είμαστε πιο, να είσαστε μάλλον πιο ειλικρινείς να πείτε ότι εδώ υπάρχουν ενεργειακά συμφέροντα και άλλου είδους συμφέροντα και αυτά εξυπηρετεί και το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να προτείνω τώρα να περιορίσουμε όλες τις παρεμβάσεις σε ένα δίλεπτο για να μπορέσουν να λάβουν όλοι το λόγο. Ο κύριος Λίσεκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Γενική Γραμματεύ. Ήσασταν πολύ συγκεκριμένος και σαφή. Θα ήθελα να θέσω τρει ερωτήσει εν συντομία. Η πρώτη αφορά αυτό που προανέφεραν και οι συνάδελφοι, δηλαδή το pooling and sharing, την FE ε, άμυνα, το smart ε, defense και μάλιστα ακούσαμε τις προάλλες ε, στην υποεπιτροπή ότι θα έχουμε 300 εκατομμύρια ευρώ ε, οικονομίες χάρη στο pooling and sharing. Ε, έγιναν ε, ε, κάτι τέτοιες αναφορές. Ε, βέβαια, έχουμε 30 δισεκατομμύρια συνολικά, οπότε πολύ, πολύ περισσότερα. Πιστεύετε ότι θα ασκήσετε πιέση στα κράτη-μέλη για να σταματήσουν τις περικοπές ε, στις αμυντικές ε, δαπάνες. Σε ό,τι αφορά την αντιπυραυλική άμυνα, υπάρχουν πολλοί ευρωσκεπτικιστές στην Ευρώπη. Πώς θέλετε να πείσετε, όχι τους πολιτικούς, πώς το ΝΑΤΟ θα πείσει τους πολίτες στην κοινή γνώμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι πρόκειται για ένα σχέδιο που θα, ε, θα προστατεύσει την Ευρώπη και δεν θα εξυπηρετήσει μόνο τα συμφέροντα των Αμερικανών, αλλά την ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για τη Γεωργία. Είμαι ο εισηγητή για την έκθεση για τη Γεωργία και θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για τα παρήγορα λόγια και τα ελπιδοφόρα που μα είπατε για την ε, Γεωργία. Σε ό,τι αφορά τη μελλοντική ε, προσχώρηση τη Γεωργία ε, στο ΝΑΤΟ, παρόλο που υποστηρίζεται από μεγάλο τμήμα τη κοινωνία τη Γεωργία και των πολιτικών κομμάτων, έχουμε πολλού πολέμιου εντό του ΝΑΤΟ που είναι και μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώ θα πείσετε τα μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να αλλάξουν τη θέση του στο ΝΑΤΟ και να δεχτούν την προσχώρηση τη Γεωργίας σε αυτό το θεσμό. Ο κύριος Βάγκελ. Äh, Ευχαριστώ. Κύριε Γενική Γραμματεύ, μου άρεσε αυτό που είπατε, ότι θα πρέπει να ε, είμαστε έτοιμοι απέναντι στο άγνωστο και στο απρόβλεπτο που θα λάβει η χώρα και που θα επηρεάσει την ασφάλειά μας. Συμφωνώ λοιπόν. Το θέμα είναι ότι το απρόβλεπτο θα πρέπει να το περιορίσουμε κάπως. Ε, σήμερα έχουμε πάρα πολλά απρόβλεπτα και ευνίδια περιστατικά, υπερβολικά πολλά θα έλεγα. Έχω λοιπόν μία ερώτηση. Θεωρείτε ότι ένας πιθανός τομέας για καλύτερη συνεργασία και καλύτερο συντονισμό μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ θα ήταν η, πρόληψη κατά κάποιο τρόπο το να προλάβουμε αυτές τις διαδικασίες και αναφέρομαι σε διαδικασίες και σχέδια που είναι μερικά προβλέψιμα και άλλα απρόβλεπτα. Σε ό,τι αφορά τα απρόβλεπτα, είδαμε ότι το ΝΑΤΟ δεν είχε και μεγάλη επιτυχία για να μην πω ότι απέτυχε κιόλα. Θεωρώ ότι τη συνεργασία μας θα πρέπει να την ενισχύσουμε, όχι μόνο εφαρμόζοντας κάποια θέματα επιμελητίας ε, και με λογιστικούς υπολογισμούς, αλλά και ε, με κάποιους εφάνταστους τρόπους. Επίσης, τι γίνεται με τη Μακεδονία, λέει ο, ο και με τη θέση της, ε, ΦΥΡΟΜ φυρών στο ΝΑΤΟ. είχαμε και την απόφαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Τι γίνεται, γιατί στην περιοχή αυτή το ΝΑΤΟ έχει σημαντική επιρροή και παρουσία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γενικός Γραμματέας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά. Καταρχήν, κύριε Βανόρντεν. Εγώ δεν είμαι ε, η για τα θεσμικά ζητήματα. Και δεν με ενδιαφέρει ποιο ακριβώ κάνει τι, ποιο είναι αρμόδιο γιατί. Εμένα με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν. Και εντοπίσαμε πολύ σημαντικέ αδυναμίε και κενά σε ό,τι αφορά τι στρατιωτικέ ικανότητε. Διδαχθήκαμε κάποια μαθήματα από τις επιχειρήσεις μας, ιδιαίτερα στο Αφγανιστάν και στη Λιβύη. Εκεί, Στη Λιβύη, εκεί πραγματικά αντιλήσαμε σημαντικά διδάγματα και εκεί εντοπίσαμε και πολύ σημαντικά κενά και αδυναμίες στις επιχειρήσεις μας. το σκοπός μας τώρα είναι να πληρώσουμε αυτά τα κενά και να διορθώσουμε αυτές τις αδυναμίες. Δεν με ενδιαφέρει αν θα γίνει αυτό στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρκεί να πληρωθούν τα κενά και να διορθωθούν τα λάθη. 21 χώρε ε, είναι μέλη και στους Και φυσικά θα πρέπει και είναι το χρέος μας απέναντι στους φορολογουμένους ε, να έχουμε αποτελεσματικό έργο γιατί έχουμε τους ίδιους φορολογούμενους και τις ίδιες στρατιωτικές ικανότητες. Χρειαζόμαστε περισσότερες επενδύσεις στις ε, μεταφορικές μας δυνατότητες. Έχουμε πολλούς στρατιώτες στην Ευρώπη, αλλά δεν μπορούμε να τους μετακινήσουμε από τη μία περιοχή στην άλλη, για να το πω ε, περιγραφικά. Επίσης, τον αέριο εφοδιασμό, το χρειαζόμαστε, το μάθαμε από την ε, σε στη Λιβύα. Χρειαζόμαστε καλύτερες ικανότητες ε, στα θέματα ε, επιτήρησης, παρακολούθησης, αναγνώρισης. Θέλουμε λοιπόν επενδύσεις στα ντρόν, σε αυτά τα μη επαδρομένα αεροσκάφη, ώστε να συγκεντρώσουμε πληροφορίες και να μπορέσουμε να καθοδηγήσουμε σωστά ε, και να λάβουμε εμπεριστατωμένα τις πολιτικές και στρατιωτικές μας αποφάσεις. Πρόκειται για σημαντικά κενά λοιπόν και αδυναμίες που έχουμε εντοπίσει. Και όπως είπα, στην διάσκεψη κορυφής του ΝΑΤΟ πέρυσι στο Σικάγο, οι σύμμαχοι και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέλαβαν τη δέσμευση να επενδύσουν στον εναέριο ανεφοδιασμό και σε τέτοιες ικανότητες. Αν θα το κάνουν αυτό μέσω της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Υπηρεσίας, γιατί όχι. Εμένα δεν με ενδιαφέρει ποιος θα το κάνει, ποια θα είναι, ποιος θα είναι ο αρμόδιος οργανισμός. Με ενδιαφέρει να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει. Και γι' αυτό συμφωνώ ότι το πιο σημαντικό που θα πρέπει να αποφασίσει το Συμβούλιο στη διάσκεψη κορυφή του Δεκεμβρίου είναι να επενδύσει επαρκή κονδύλια σε στρατηγικές ικανότητες που τις χρειαζόμαστε διακαώς. Αυτή θα είναι η πιο σημαντική απόφαση που θα πρέπει να ληφθεί το Δεκέμβριο. Κυρία Κρόμπερκ, με ρωτήσατε κατά πόσο το ΝΑΤΟ θα αναλάβει ρόλο στο Ιράν ή σκοπεύει να κάνει κάτι τέτοιο. Όχι. Κατηγορηματικά λέω όχι. Ουδέποτε δεν έκανα σχετικέ δηλώσει. Το αντίθετο. Και θα ήθελα να πω ότι το ΝΑΤΟ, η Βορειοατλαντική Συμμαχία, δεν έχει εμπλακεί σε θέματα του Ιράν. Και στηρίζουμε τι διεθνεί προσπάθειε να αναβρεθεί μια πολιτική και διπλωματική λύση στο Ιράν. Σε ό,τι αφορά την αντιπυραυλική άμυνα. Με ρωτήσατε κατά πόσο η αλλαγή της προσέγγισης σε φάσεις θα μπορούσε να βελτιώσει τη στενότερη συνεργασία με την Ρωσία για τα θέματα αντιπυραυλικής άμυνας. Πολύ σημαντική η ερώτηση και εύστοχη και η απάντησή μου είναι ναι, θα έπρεπε να βελτιωθεί αυτή η συνεργασία. Γιατί μέχρι στιγμής οι ανησυχίες της Ρωσίας αφορούσαν κυρίως την τέταρτη φάση, η οποία κυρώθηκε. Και τώρα, μια και είδαμε ότι ακυρώθηκε, de facto δεν έχουν λόγο οι ρωσικές ανησυχίες. Οπότε αν υπάρχει πολιτική βούληση στη Μόσχα για συνεργασία, θεωρώ ότι με την ακύρωση της τέταρτης φάσης διανοίγεται ο δρόμος για μια συμφωνία με θέμα το πώς θα μπορούσαν να συνεργαστούν το ΝΑΤΟ και η Ρωσία σε θέματα αντιπυραυλικής άμυνας. Επιπλέον θα ήθελα να πω ότι το γεγονός ότι τέταρτη και τελευταία φάση έχει καταργηθεί, δεν αλλάζει το γεγονός ότι ολόκληρος ο πληθυσμός των κρατών του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλύπτονται από το αντιπυραυλικό σύστημα του ΝΑΤΟ. Γιατί οι πρώτες τρεις φάσεις θα εφαρμοστούν με βάση το σχέδιο και θα καλύψουν ολόκληρο τον πληθυσμό των κρατών του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς τον κύριο Αγκουράκη. Κοιτάξτε, ρωτήσατε πότε θα πάψει πλέον να υπάρχει η κατοχή του πεδίου, μεταξύ άλλων. Ε, το πιο ενδιαφέρον από όλα είναι το εξής, ότι στην περιοχή οι πολίτες, οι άνθρωποι δεν θεωρούν ότι είναι υποκατοχή των αντίον. Πρόσφατα, όταν η Κάθη ε, Άστον ολοκλήρωσε αυτή τη συμφωνία μεταξύ του Βελιγραδίου και της Πρίστινα και οι δύο πλευρές ζήτησαν από τον ΝΑΤΟ να παραμείνει εκεί και να εγγυάται το ΝΑΤΟ την εφαρμογή της συμφωνίας. Άρα δηλαδή δεν μπορούμε να μιλάμε για κατοχή. Βεβαίως ε, χαίρομαι που το ΝΑΤΟ τελικά αντιμετωπίζεται ως ένας ε, ε, αμερόληπτος εγγυητής της ειρήνης και της αθερότητας. Εγώ μπορώ να σας πω ότι θα παραμείνουμε μέχρι να ολοκληρωθεί η εντολή των Ηνωμένων Εθνών. Αυτή είναι η εντολή που μας έχει δοθεί και είναι υποχρέωσή μας να την εφαρμόζουμε την εντολή αυτή. Να διασφαλίζουμε την ε, ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών. Επίσης με ρωτήσατε σχετικά με το Αφγανιστάν. Μα νομίζω υπάρχει ένας ε, σαφής χαρτής ε, πορείας. Μέχρι το τέλος του 2014 η δική μας η αποστολή θα έχει ολοκληρωθεί. Θα παραμείνουμε βέβαια και με το, μετά το 2014 όχι με μάχημες δυνάμεις αλλά με δυνάμεις ε, εκπαίδευσης για να βοηθήσουμε τις ε, τοπικές ε, δυνάμεις του Αφγανιστάν. Κυρία Λισμπερτ, με ρωτήσατε αν θα κάνουμε κάτι για να περιορίσουμε τις περικοπές τους αμυντικούς προπολογισμού. Όπως ξέρετε, το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να παρέμβει σε κάτι τέτοιο. Αυτό είναι θέμα εθνικής απόφασης. Για μας λοιπόν υπάρχει ένα πρόγραμμα και με βάση αυτό ε, τα μέλη του ΝΑΤΟ έχουν αναφέρει ότι οι σύμμαχοι που δαπανούν πάνω από 2% σε αμυντικούς ε, προϋπολογισμούς, γιατί υπάρχει αυτή η δέσμευση του 2%, αυτή είναι εντάξει. Οι άλλοι που είναι κάτω από το 2% θα προσπαθήσουν να φτάσουν στο 2%. Αυτό βέβαια δεν είναι νομική, νομικός όρος, είναι ε, πολιτική αν θέλετε υποχρέωση. Και οποτεδήποτε ε, επισκέπτομαι τις πρωτεύουσες των κρατών μελών και σύντομα θα πάω στη Βαρσοβία, επαναλαμβάνω αυτό που σας είπα. Επίσης, να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε διεξάγει τον πολιτικό διάλογο με κυβερνήσεις αλλά και με ε, βουλευτές και έχω διαπιστώσει θετική αντίδραση. Και μπορώ να σας αναφέρω μια χώρα όπου τα βασικά πολιτικά κόμματα κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία και με βάση αυτή σιγά σιγά ε, θα πλησιάσουν το 2%. Γι' αυτό λοιπόν για ένα γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ είναι σημαντικό να έρχεται σε άμεση επαφή με κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους γιατί εδώ γίνεται λόγος για αμυντικούς προϋπολογισμούς και γενικότερα βέβαια για ε, πολιτικές εξυγίανσης ε, των οικονομικών. Επίσης με ρωτήσατε πώς μπορούμε να πείσουμε τους ανθρώπους ότι όλα αυτά είναι και προς όφελος των Ευρωπαίων. Νομίζω είναι σαφές ότι αντιμετωπίζουμε πυραυλική απειλή. Πάνω από 30 χώρες έχουν αποκτήσει την ε, τεχνική αυτή ώστε να μπορούν να πλήξουν στόχους στην Ευρώπη. Άρα δηλαδή είναι προς όφελος της Ευρώπης να αναπτύξει και αυτή ένα σύστημα Άμυνα και προστασίας από αυτή την πυραυλική απειλή. Όσον αφορά τώρα τη Γεωργία, κοιτάξτε, η απόφαση που πήραμε στο Βουκουρέστι το 10 ε, στη συνάντηση κορυφή του ΝΑΤΟ εξακολουθεί να ισχύει. Είπαμε ότι η Γεωργία θα γίνει μέλος του ΝΑΤΟ υπό την προπόθεση ότι θα τηρεί τους όρους. Και έχουμε συστήσει μια ειδική επιτροπή ΝΑΤΟ Γεωργίας. Εκεί λοιπόν συνεργαζόμαστε να προχωρήσει η υπόθεση και η Γεωργία να συνεχίσει και αυτή τις ε, μεταρρυθμίσεις της με τελικό στόχο κάποια μέρα στο πότερο μέλλον να προσχωρήσει στο ΝΑΤΟ. Δεν ε, έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο, υπολείπονται ακόμα πολλά, αλλά ε, νομίζω ότι η νέα, η κυβέρνηση του, της Γεωργίας έχει επαναλάβει τις ε, φιλοδοξίες που είναι αυτές που σας παρουσίασα. Άρα δηλαδή εναπόκειται πλέον στη Γεωργία αυτή να εκπληρώσει τους όρους. Ε, τέλος ο κ. Μπόγγελ με, μου έκανε μια ερώτηση σχετικά με τη μελλοντική διεύρυνση. Ε, εμείς έχουμε επαφές με τα Σκόπια. Ε, έχουμε δραστηριοποιήσει τις επαφές και το 8 επίσης Βουκουρέστη Βουκουρέστι αποφασίσαμε ότι θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσει 11 με τα Σκόπια τη στιγμή που θα έχει εξευρεθεί μια αμοιβαίω αποδεκτή λύση στο θέμα του ονόματος, της ονομασίας της χώρας. Η χώρα το γνωρίζει, οι Σκοπιανοί το γνωρίζουν. Έτσι λοιπόν εμείς από πλευρά ΝΑΤΟ έχουμε κάνει ό,τι μπορούσαμε. Αμέσως θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις μόλις βρεθεί λύση στο θέμα της ονομασίας. Γι' αυτό λοιπόν εγώ ενθαρρύνω όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να μην φυστούν κόπου για να βρουν κάποια λύση σε αυτό το πρόβλημα. Κατά την άποψή μου είναι εφικτό κάτι τέτοιο. Μπορεί να υπάρξει εάν υπάρχει πολιτική βούληση. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς λέει ο Πρόεδρος. Τέσσερα ονόματα έχω, ή τρία αν θέλετε, ε, είχα αρχικά στον κατάλογο, ε, τώρα έχουν προσθεθεί άλλοι τρεις, φτάσαμε στους έξι εσείως, αν όμως τελικά ο καθένας μιλήσει για ένα περίπου λεπτό, ίσως και να τα καταφέρουμε. Η Βερονίκ, είστε η πρώτη. Merci, Monsieur le Président. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ράσμουσεν, μία ερώτηση έχω μόνο. Το ΝΑΤΟ γνώρισε τις επιθέσεις και τους φοβαρδισμούς του Ισραήλ στη Δαμασκό και κάνατε κάποιο συντονισμό των επιχειρήσεων και σας θέτω την ερώτηση γιατί στις 7 Μαρτίου 2013 το ΝΑΤΟ υπέγραψε Συμφωνία εταιρική Σχέσης και Συνεργασίας με το Ισραήλ. Διμερή συμφωνία. Και μάλιστα διαβάζαμε τότε στον τύπο το Ισραήλ γίνεται de facto μέλος του ΝΑΤΟ. Η εταιρική αυτή σχέση θα βελτίωνε τη διαδικασία θετικού σχεδιασμού μεταξύ της Ευρωπαϊκής, των Ηνωμένων Πολιτειών, συγγνώμη, του ΝΑΤΟ και του Ισραήλ σε σχέση με οποιασδήποτε μελλοντικέ επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Αυτά προέβλεπε η συμφωνία. Δύο μήνες ε, πριν τις σημερινέ επιχειρήσεις. Δύσκολο κανείς θα πιστεύω ότι δεν έγινε, ε, έγιναν αυτέ οι επιχειρήσει χωρίς κανένα συντονισμό. Πώς αναλύεται εσεί και πώς χαρακτηρίζεται αυτή την επιχείρηση. Η κυρία Σχάκε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Γενική Γραμματέα. Μιλήσατε για την ανάγκη ηγεσία αυτών των με των βαλόμενων κόσμο και ε, την ανάγκη για ικανότητες, ε, χωρίς τι οποίες είναι κενή η πολιτική ηγεσία. Τι γίνεται για τον κυβερνοχώρο σε ό,τι αφορά τις τεχνολογίες και την άμυνα. Στη ΣΥΠΑ διαπιστώθηκε ότι χρειάζονται σχετικές ε, επιθετικέ ικανότητε, ικανότητες. Διάβασα το σχετικό εγχειρίδιο Πώς θα διασφαλίσετε ότι η ελευθερία και η ασφάλεια και στο θέμα της τεχνολογίας θα διασφαλιστούν. Ένα τελευταίο ερώτημα για την Συρία, όπου θεωρώ ότι πλέον χρειάζονται ε, ισχυρά μέτρα. Παρακολούθησα το θέμα αυτό πολύ προσεκτικά τα τελευταία χρόνια και σε διάφορες περιστάσεις αναφέρατε από μόνο σας ότι το ΝΑΤΟ δεν πρόκειται να εμπλακεί στη Συρία. Σας ρωτώ λοιπόν γιατί. Mr. Ruzek. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μόλις επέστρεψα από τα Βαλκάνια, κύριε Ρούτσεκ. Μιλώντας λοιπόν για τα Βαλκάνια, έχουμε αφήσει ανοιχτές κάποιες δουλειές εκεί σε ό,τι αφορά τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ. Η Φύρο Μακεδονία αναφέρθηκε, λέει ο μιλητής. Τι γίνεται όμως με χώρες όπως το Μαυροβούνιο, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Σερβία. Ποιε θεωρείτε ότι είναι οι προοπτικέ των χωρών αυτών. Στην επόμενη διάσκεψη του ΝΑΤΟ θα γίνει διεύρυνση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπιτικόφερ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Γενικά, Γενική Γραμματέα, τρεις ερωτήσεις. Το ΝΑΤΟ τι θεωρείτε ότι θα πρέπει να κάνει για να προωθήσει τον πυρηνικό αφοπλισμό. Δεύτερο ερώτημα. στην ε, Ανατολική Ασία γίνεται μια κούρσα εξοπλισμών, την οποία και τροφοδοτούμε εμείς. Ποια η άποψή σας επ' αυτού. Θα πρέπει να δείξουμε μεγαλύτερη σύνεση σε ό,τι αφορά την πολιτική μας, σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές στην περιοχή αυτή. Και τρίτον, πέρα από τα θέματα αντιπρευλικής προστασίας, ποια θεωρείτε ότι είναι η κορυφαία μας προτεραιότητα ως Ευρωπαίοι και εσείς ως ΝΑΤΟ σε ό,τι αφορά την συνεργασία για θέματα άμυνας με τη Ρωσία. Και στο πλαίσιο αυτό είμαι βέβαιος ότι είδατε την έκθεση τεσσάρων πρώην ε, ε, ηγετών για την αμοιβαία ε, εμπιστοσύνη σε θέματα διακρατική προστασίας. Ποια είναι η άποψή σας από αυτόν, ο κύριος Κυρίλοφ. Ναι, όπως ξέρετε πέρσι έγινε στον Μπούργκας μια επίθεση, μια τρομοκρατική επίθεση μεγάλης κλίμακας σε ευρωπαϊκή Επικρέτεια. Και μετά από αυτή έγιναν πολλές συντονισμένες έρευνες ασφαλώς, οι οποίες προς το παρόν έχουν καταλήξει σε αντιέξοδο. Οι ΗΠΑ θεωρούν ότι έδρασε η Χεσμολά και πιέζουν τους εταίρους τους να αντιμετωπίσουν το θέμα της Χεσμολά επισήμως. Αφετέρου υπάρχει ακόμα Υπάρχουν κάποια ερωτηματικά. Ασφαλώς αυτό δεν αποτελεί θέμα βασικό δικό σας, αλλά ασφαλώς και θα έχει συζητηθεί. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την τελευταία αυτή επίθεση της Χεσμολά, σχετίζεται ενδεχομένως με ενδεχόμενη δράση στο Ιράν, την οποία και απέφχομαι. Θα πρέπει λοιπόν ενδεχομένως πριν δράσουμε στο Ιράν να αντιμετωπίσουμε το θέμα της Χεσμολά. Tack så mycket, herr ordförande. Två mycket Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, η Γαλλία ανέλαβε κάποια δράση στο Μάλι. Τι γίνεται με το ΝΑΤΟ. Τι γίνεται με τα ρωσικά αεροσκάφη που πέρασαν ε, σχεδόν κοντά από τα σουηδικά σύνορα. Και αν ήταν χώρα του ΝΑΤΟ θα συνέβαινε κάτι τέτοιο. Ποιες είναι οι δικές εκτιμήσεις. Σας ευχαριστώ τώρα ο κύριος Ράσμουσεν για να απαντήσει. Σας ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα να απαντήσω στην κυρία Δεκάιζερ. με ρωτήσατε κατά πόσο το ΝΑΤΟ συντόνισε με το Ισραήλ τις επιχειρήσεις, της, ε, την επιδρομή της βομβαρδισμού. Ε, Σας απαντώ κατηγορηματικά όχι. Ναι μεν έχουμε εταιρική σχέση με το Ισραήλ και έχουμε και την εταιρική σχέση που αποκαλούμε μεσογειακό διάλογο. Και ο διάλογος αυτός δεν περιορίζεται μόνο στο Ισραήλ, αλλά και σε έξι άλλε χώρε τη Βορειοαφρική και τη Μέση Ανατολή. Και έχουμε προγράμματα στρατηγική συνεργασία με όλε αυτέ τι χώρε. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν συντονίσαμε την, τις επιθέσεις, τις επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Σύρια. Κύριε Χάκε, μιλήσατε για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Σίγουρα αυτό το θέμα είναι από τις σημαντικότερες ε, καινοφανείς απειλές για την ασφάλεια και θα πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Και μάλιστα στο ΝΑΤΟ ε, προσπαθούμε να ενισχύσουμε την ε, άμυνά μας στον κυβέρνο χώρο και το πρώτο μας βήμα ήταν η ενίσχυση της άμυνας των δικτύων μας του ΝΑΤΟ των εταιρικών δικτύων και το χρειαζόμαστε αυτό γιατί πολύ τακτικά υφιστάμεθα επιθέσεις κάτι που δεν μας ευνηδιάζει βέβαια. Μέχρι στιγμής ε, καταφέραμε με ιδιαίτερη επιτυχία να προσπίσουμε τα συστήματά μας, τα ανατοικά συστήματα και αυτό είναι το πρώτο βήμα. Στη συνέχεια θα πρέπει να εξετάσουμε κατά πόσο και με ποιον τρόπο θα αναπτύξουμε μια ικανότητα που θα βοηθήσει τους μεμονωμένους μας ε, συμμάχους ε, όταν βάλλονται από τέτοιες επιθέσεις. Γιατί μερικοί σύμμαχοι μπορούν να αυτοπροστατευτούν κατά τέτοιων ε, κυβερνοεπιθέσεων, αλλά άλλοι σύμμαχοι θα ήθελαν πολύ το ΝΑΤΟ να έχει την ικανότητα να τους προστατεύσει. Ένα είδος ομάδας άμεσης δράσης που θα μπορούσε με αίτημα της ε, πληττόμενης χώρας να αναλάβει δράση για να αποτρέψει τέτοια επίθεση στον κυβερνοχώρο. Είναι από τα στοιχεία λοιπόν που επεξεργαζόμαστε και σίγουρα η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο είναι ένα θέμα για το οποίο χρειαζόμαστε στενή συνεργασία και με τους εταίρους παγκοσμίω, γιατί η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο είναι ένα πραγματικά διασυνοριακό θέμα παγκόσμιο και πιστεύω ότι θα πρέπει να τεθεί σε, στις συζητήσεις μας με χώρες που εστερνίζονται αυτές τις απόψεις. Τώρα, με ρωτήσατε για τη Συρία. Γιατί, λέτε, το ΝΑΤΟ δεν έχει καν την πρόθεση να επέμβει στρατιωτικά στη Συρία. Και πολύ συχνά ακούω αυτή την ερώτηση. Γιατί επικαλούνται τις επιτυχείς επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ στη Λιβύη και ρωτάνε γιατί δεν κάνετε το ίδιο και στη Συρία. Υπάρχει σαφέστατη όμως διαφορά μεταξύ Λιβύης και Συρίας. Στη, Λιβύα, στη Λιβύη συγγνώμη, είχαμε σαφή και απερίφραστη εντολή του ΟΗΕ για να προστατεύσουμε τους άμαχους, τον άμαχο πληθυσμό και είχαμε και την α, θερμή υποστήριξη και την ενεργό υποστήριξη των γειτονικών χωρών. Δεν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, αντίστοιχες προϋποθέσεις στην περίπτωση της Συρίας. Στη Συρία η κοινωνία είναι πολύ πιο περίπλοκη. Η κατάσταση είναι πολύ σύνθετη. Και θεωρώ ότι μια εξωτερική στρατική παρέμβαση ίσως έχει απρόβλεπτες επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή. Στην συγκεκριμένη περίπτωση θεωρώ ότι η κατάλληλη λύση είναι πολιτική. Πάντως συμμερίζομαι πλήρως την ε, απογοήτευση και τη ματέωση που νιώθουμε βλέποντας ανήμποροι την αποτρόπαια κατάσταση στη Συρία. Και πραγματικά ε, επήγει το θέμα. Θα πρέπει κατεπηγόντως ε, η διεθνή κοινότητα να στείλει ένα ισχυρό, κατηγορηματικό και ενιαίο μήνυμα προς το καθεστώς της Δαμασκού. Μέχρι στιγμής το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ δεν κατάφερε να καταλήξει συνένεση και λυπούμε ειλικρινά γι' αυτό γιατί θεωρώ ότι έχουμε ένα πολιτικό πλαίσιο που θα μπορούσαμε να το, χρησιμοποιήσαμε, να το χρησιμοποιήσουμε. Όπως θα θυμάστε, τον Ιούνιο του 2012 η ομάδα δράσης για τη Συρία εξέδωσε μια διακήρυξη που τη συνυπέγραψε όλα τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΕ. Και στη δήλωση αυτή, στη διακήρυξη αυτή, αναφέρεται σαφώς ότι το καθεστώς του Δαμασκού, της Δαμασκού θα πρέπει να ξεκινήσει μια διαδικασία μετάβασης προκειμένου να υλοποιηθούν οι εύλογες ε, προσδοκίες και βλέψεις του Συριακού λαού. Θεωρώ λοιπόν ότι μια πολιτική λύση θα μπορούσε να βασίζεται σε αυτή τη διακήρυξη. Φυσικά για κάτι τέτοιο χρειαζόμαστε ένα ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Τώρα, κύριε Ρόουτσεκ, με ρωτήσατε για τις α, ενταξιακές προοπτικές των βαλκανικών χωρών. Το Μαυροβούνιο, το Μοντενέγρο, ε, επιτέλεσε σημαντική πρόοδο. Γι' αυτό και έχουμε ένα σχέδιο δράσης ένταξης για το Μοντενέγκρο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν εκπληρωθεί όλες οι προϋποθέσεις, αλλά πραγματικά έχω μείνει εντυπωσιασμένος από την πρόοδο και το έργο που επιτελεί ε, το Μαυροβούνιο. Τώρα, Βοσνία και Ριζεγοβίνη. Εκεί έχουμε μια πολιτική στασιμότητα, μια πολιτική αποτελμάτωση. Πριν από λίγα χρόνια είχαμε θέσει κάποιου όρου ε, για το σχέδιο δράση ένταξη τη Βοσνία Ερζεγοβίνη και δηλώσαμε ότι είμαστε πρόθυμοι να ενεργοποιήσουμε αυτό το σχέδιο δράση ένταξη τη Βοσνία από τη στιγμή που οι Βόσνοι υλοποιήσουν κάποιες ε, σχετικά μετριοπαθείς ε, ε, μεταρρυθμίσεις σε ό,τι αφορά την κυριότητα σε θέματα άμυνας. Και μάλιστα μου είπαν οι ηγέτες στη Βοσνία ότι είναι πρόθυμοι να υλοποιήσουν την πολιτική συμφωνία του περασμένου έτους, αλλά μέχρι στιγμής πρόοδος δεν έχει γίνει και είναι κρίμα. Αν η Βοσνία υλοποιήσει τις υποχρεώσεις της, εμείς είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε αμέσως. Και σε ό,τι αφορά τα Σκόπια, νομίζω ότι απάντησα. Δεν θεωρώ ότι η πρόσφατη πολιτική συμφωνία Βελιγραδίου-Πρίστινας που βελτιώνει και διευκολύνει την πρόοδο σε ό,τι αφορά την ενταξιακή διαδικασία των Δυτικών Βαλκανίων στις ευρωατλαντικές δομές πρέπει να μεληθεί. Εναπόκειται στις χώρες αυτές να υλοποιήσουν τις υποχρεώσεις. Αν το κάνουν εμείς είμαστε έτοιμοι, πανέτοιμοι. Και θα είμαστε ε, πανέτοιμοι όταν και εκείνοι δηλώσουν τη δική τους ετοιμότητα. Τώρα, αν θα είναι η επόμενη διάσκεψη κορυφή, ε, ενταξιακή διάσκεψη, διάσκεψη της διεύρυνση. Δεν έχουμε αποφασίσει πότε θα γίνει η επόμενη διάσκεψη κορυφή. Και για να γίνει κανεί μέλος του ΝΑΤΟ θα πρέπει να πληρεί κάποια κριτήρια και προϋποθέσεις. Εναπόκειται στι υποψήφιες χώρε να εκπληρώσουν αυτέ τι προποθέσει και τα κριτήρια. Κύριε Βουτικόφερ, ζητήσατε πυρηνικό αφοπλισμό. έχουμε θετήσει ένα στρατηγικό δόγμα και σε αυτό το, αυτή τη στρατηγική του ΝΑΤΟ επανεπιβεβαιώνουμε και διατρανώνουμε αυτό που υποστηρίζουν ήδη από το 1970 πολλές χώρες διεθνώς ότι στόχος μας είναι ένας κόσμος απαλλαγμένος από τα πυρηνικά όπλα. Αυτό είναι το μεγαλεπίβολο όραμα που συμμεριζόμαστε οι περισσότεροι. Αλλά αφελείς δεν είμαστε. Δηλώσαμε ότι στο μέτρο που υπάρχουν πυρηνικά, το ΝΑΤΟ θα παραμείνει και πυρηνική συμμαχία. Μακάρι όμως ε, να μειωθούν ε, τα πυρηνικά όπλα και με ισορροπημένο τρόπο. Και εδώ οφείλω να πω ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ έχουν μειώσει τον αριθμό ε, των πυρηνικών τους όπλων και μάλιστα αισθητά από το τέλος του ψυχροπολέμου. Κάτι που δεν ισχύει για τη Ρωσία. Γι' αυτό τονίζω ότι ναι, μεν είμαστε υπέρ της, του περιορισμού των πυρηνικών όπλων, αλλά με ισορροπημένο τρόπο. Και για την ευρωατλαντική ασφάλεια διάβασα την έκθεση της ομάδας Kissinger με μεγάλο ενδιαφέρον και σίγουρα χρειαζόμαστε μία δέσμευση και της Ρωσίας και προσκαλέσαμε τη Ρωσία να συνεργαστεί μαζί μας σε θέματα αντιπυραυλικής άμυνας και έχουμε σημειώσει πρόοδο σε πολλά θέματα συνεργασίας αλλά σίγουρα θα είναι λιδία αλήθως και το θέμα της αντιπυραυλικής άμυνας. Μέχρι στιγμή δεν έκανε δεκτή την πρόσκλησή μα η Μόσχα. δυστυχώ επαναλαμβάνω. Αλλά εμεί θα συνεχίσουμε το διάλογό μας. Κύριε Σβένσον, με ρωτήσατε κατά πόσο αυτό το περιστατικό αυτό το επεισόδιο θα είχε λάβει χώρα αν η Σουηδία ήταν μέλος του ΝΑΤΟ. Δεν το γνωρίζω, κύριε Σβένσον. Ούτε πρόκειται να επέμβεδω στην εσωτερική συζήτηση της Σουηδίας για το ΝΑΤΟ. Παρακολούθησα αυτή την ε, συζήτηση στο εσωτερικό της Σουηδίας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αλλά επαναλαμβάνω αυτό που είπα και στη Σουηδία, ότι υπάρχει σαφής διαφορά μεταξύ του να είναι κανείς μέλος του ΝΑΤΟ και να, του να, μην είναι, του να καλύπτεται από το άρθρο 5. Για να καλύπτεται το, το άρθρο 5, ένα κράτος θα πρέπει να είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Πάντως εκτιμούμε ιδιαίτερω την πολύ στενή εταιρική σχέση που έχουμε με τη Σουηδία. Herzlichen Dank, Herr Generalsekretär. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Γενική Γραμματέα για όλα αυτά που μας είπατε. Κοιτάξτε, πρέπει να τελειώσουμε τώρα, γιατί έχει έρθει ο επόμενος ομιλητής. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γενικό Γραμματέα που μας ε, επισκέφθηκε και νομίζω ότι ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ μέχρι τη συνάντηση κορυφής ε, θα πρέπει να υπάρξουν και άλλες συζητήσεις γιατί η συνέργεια μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από την ευρωπαϊκή συνεργασία αλλά και για να υπάρχει μια σαφής γραμμή, να υπάρχει συμπληρωματική συνεργασία ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Μήπως μπορείτε σας παρακαλώ να παραμείνετε καθισμένοι μέχρι να ολοκληρώσουμε και αυτό το σημείο της μερίσιας διάταξης. Ωραία. Και όλα αυτά είναι επιγόντως απαραίτητα γιατί μπορεί να γίνουν σημαντικές αλλαγές στην Αμερικανική πολιτική. Δεν ξέρω ποια θα είναι στο μέλλον η πολιτική της Αμερικής ε, στη Μέση Ανατολή όταν θα είναι πλέον αυτάρκης ενεργειακά οι Ηνωμένε Πολιτείε. Ενδέχεται αυτό να οδηγήσει σε μετατόπιση ε, των συμφερόντων, κάτι που οπωσδήποτε θα παίξει και ρόλο στη σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΝΑΤΟ και Ηνωμένων Πολιτειών. Άρα δηλαδή είναι σημαντικό να ε, συνεχιστεί η συνεργασία. Σας ευχαριστώ θερμά για το ότι είχαμε τη σημερινή συζήτηση, αλλά πρέπει να σας πω και το εξής. Μερικές φορές, όσον αφορά τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Αμερικανούς φίλους μας, πρέπει να μην ξεχνάμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με την μη στρατιωτική της βοήθεια συμβάλλει τα μάλα ε, στην κατανομή των εργασιών. Γιατί μόνο από τον προπολισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για προληπτική πολιτική ε, εκτός Ευρώπης δίνεται περισσότερα χρήματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταβάλουν το 60% της αναπτυξιακής βοήθειας σε αυτόν τον κόσμο. Αυτό λοιπόν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στο πλαίσιο του περίφημου burden sharing. Ε, βεβαίως Παρ' όλα αυτά θέλω να πω ότι η συνεργασία πρέπει να συσφιχτεί περαιτέρω και οι Ευρωπαίοι πρέπει να έχουν περισσότερες δυνατότητες να ανταποκρίνονται στις ε, στρατιωτικές τους υποχρώσεις. Κατόπιν τούτου χαίρομαι και εγώ πάρα πολύ που θα μπορέσουμε το καλοκαίρι και το φθινόπωρο να συνεργαστούμε για να προετοιμάσουμε τη συνάντηση κορυφή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε να μας επισκεφτείτε.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 Κύριε καθίστε αν θέλετε. Τις τελευταίες ε, μέρες έχουν τεθεί κάποιες ερωτήσεις, επερωτήσεις. Μάλλον μου έχουν ζητήσει συνάδελφοι να γίνουν συντηγητές για το Ιράκ και μετά θα μπορούσαν, θα μπορούσαν να γίνουν και οι Υπουργοί ε, Άμυνας, ε, εφόσον θα είχαν διατελέσει ε, μέλη της Επιτροπής ε, Καλώς ορίζω λοιπόν τον Μάουρο Μάριο και τον συγχαίρω για την θέση του ε, ως Υπουργό Άμυνας της Ιταλίας. Σε κάποιες ε, περιπτώσεις ε, μας προκαλούν έκπληξη η επιλογή προσωπικού της Ιταλίας, γιατί ίσως είναι διαφορετικές οι διαδικασίες, αλλά σε πολλές περιπτώσεις τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ καλά. Και θεωρώ ότι στο Μάριο Μάουρο έχουμε έναν πολύ άξιο συνάδελφο στη θέση αυτή. Σας συγχαίρω. Μάριο, να μας κάνεις μια μικρή εισαγωγή προκειμένου να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Αν υπάρχει ένας ε, λόγος που λατρεύω το ότι είμαι Ιταλός, είναι ότι η χώρα μου δεν πάβει ποτέ να με εκπλήσει και ένα γεγονός που μας εκπλήσει όλους είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα ο πιο ειρηνικός άνθρωπος από την Ιταλική Αντιπροσωπεία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έγινε ακριβώ υπουργό Άμυνα. Και τέλος πάντων αυτό ήρθα εδώ να σας πω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι δηλαδή αισθάνομαι δεσμευμένος ε, και ε, στρατευμένος ε, σε πολιτικές άμυνας, οι οποίες όμως διακατέχονται από την έννοια της ασφάλειας, όχι απλά και μόνο ως ασφάλεια χωρίς να υπάρχουν προκλήσεις. Εγώ πιστεύω ότι η μεγάλη πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε μέχρι το Δεκέμβρη, η μεγάλη αυτή πρόκληση είναι να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε κατά πόσο μπορούμε να έχουμε μια τέτοια πολιτική άμυνας που θα μας επιτρέπει να προχωρήσουμε στην διαδικασία της πολιτικής ολοκλήρωσης. Η συζήτηση λοιπόν αυτή έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και αφορά το κοινό όραμα της ε, άμυνας. Ε, πρόκειται για έναν πυλώνα που μας ε, επιτρέπει να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση της ε, ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η η τελική κυβέρνηση που πρόκειψε από τις τελευταίες εκλογές τόσο δύσκολες για τη χώρα μου. Η νέα λοιπόν κυβέρνηση έχει επανδρωθεί όχι μόνο από φιλοευρωπαϊστές αλλά τα έλεγα και με μια πεντεραλιστική σφραγίδα, κάτι το οποίο μεσοπρόθεσμα θα επηρεάσει τις αποφάσεις που θα ληφθούν θέσεις που θα παρουσιαστούν προς όφελος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγώ έμαθα ότι υπάρχει η δυνατότητα με αξιοπρέπεια να βιώνει κανείς ε, τις ε, ευρωπαϊκές εξελίξεις ε, και αυτό, επιτρέψτε μου να επαναλάβω, Επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω ότι αυτή είναι και η θέση την οποία πρόκειται να λάβει η Ιταλική κυβέρνηση κατά τους επόμενους μήνες και χρόνια. Αυτή είναι μια θέση η οποία θα επικεντρώνεται ακριβώς στο τι είναι απαραίτητο να προχωρήσει η διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο θεωρώ ότι χωρίς πολλά λόγια πρέπει κανείς να αντιμετωπίσει τα προβλήματα, να δει τι είναι εκείνο το οποίο αναχαιτίζει ακριβώς αυτό το κοινό όραμα της άμυνας. Καλούμεθα να εντοπίσουμε τα προβλήματα, να βρούμε λύσεις που να είναι συνεπείς με τις αξίες μας, λύσεις οι οποίες αποτελούν και το γενετικό κώδικα του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Εγώ δεν απεκδίωμαι των ευθυνών μου. Πιστεύω ότι σήμερα η πολιτική άμυνα στην Ευρώπη υποφέρει από δύο βασικά προβλήματα. Το πρώτο έχει σχέση με την επιβράδυνση της ε, διαδικασίας ε, σύσφυξης ε, των σχέσεων στον τομέα της άμυνας ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Έχω λοιπόν την εντύπωση ότι σήμερα η διαδικασία αυτή επιβραδύνεται κυρίως ε, λόγω της στάσης ε, των ε, κρατών μελών δεν υπάρχει πλέον τόσο μεγάλη θέληση για κοινέ απόψεις. Δεν λέω ότι έχει υπάρξει πλήρης αναχέτηση αυτής της διαδικασίας, αλλά παρόλα αυτά πιστεύω ότι τα ευρωπαϊκά κράτη πρέπει να προχωρήσουν με μεγαλύτερο ρυθμό προς την κατεύθυνση επίτευξης του στόχου που θα είναι μια ευρωπαϊκή άμυνα σταθερή και ολοκληρωμένη. Γνωρίζουμε ότι έχουν ληφθεί πάρα πολλές πρωτοβουλίες ε, πρωτοβουλίες ε, για να βελτιωθούν όσα έχουν επιτευχθεί ή για να υπάρχει καλύτερη λειτουργία. Εγώ όμως νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε περαιτέρω, δηλαδή να επανέλθουμε στον ενθουσιασμό που υπήρχε στο πρόσφατο παρελθόν για την πολιτική άμυνας και ασφάλειας. Και επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω τη φάση εκείνη ε, όταν πρωτοήρθα και εγώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περίπου το 2000 όταν δηλαδή η Ευρώπη ε, διοχέτευε τους σωστούς πόρους ε, και όχι μόνο χρήματα, δεν μιλώ μόνο για χρήματα αλλά και πνευματικούς και άλλους πόρους προς την κατεύθυνση της εξωτερικής πολιτικής ασφάλειας. Μπορέσαμε λοιπόν να επεξεργαστούμε μια τέτοια στρατηγική η οποία να υπηρετεί τους βασικούς στόχους από στρατιωτικού δυναμικού μπορέσαμε ε, σιγά σιγά να αναπτύξουμε περαιτέρω τις δυνατότητές μας μέσα σε ένα κοινό πλαίσιο και είμαι πεπισμένος ότι όλα αυτά ήταν ιδιαίτερα θετικά. Όχι μόνο για την πολιτική ασφάλειας και άμυνας, αλλά γενικότερα για την Ευρώπη, στο σύνολό της. Και επιπλέον είμαι πεπισμένος ότι μπορούμε να ανακτήσουμε αυτή τη ε, δυνατότητα να κάνουμε προβλέψεις για το μέλλον. Γιατί μην ξεχνάτε ότι υπήρχαν και εποχές όπου μιλάγαμε για το κοινό σύνταγμα. Οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να είναι συμβατή και με το ρόλο που θέλουμε να διαδραματίσουμε σε διεθνή διεθνές επίπεδο. Κατά την άποψή μου είναι πολύ σημαντικός ε, και ο ρόλος που μπορεί να παίξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, έτσι εδώ, μην ξεχνάμε, προκύπτουν οι επιλογές που καθιστούν την Ευρώπη ισχυρή. Και όλα αυτά πρέπει να ισχύουν και για ένα καθοριστικό τομέα που είναι ο τομέας της άμυνας. Εγώ λοιπόν εύχομαι ότι και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ε, υπάρξει συνειδητοποίηση του ότι είναι απαραίτητο να επανέλθει, να ανακάμψει αυτή η διαδικασία της εκείνης του εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής άμυνας από εδώ, από το Κοινοβούλιο, να δοθεί όθηση στα κράτη-μέλη για να λάβουν σημαντικές αποφάσεις. Το δεύτερο πρόβλημα που υπάρχει κατά την άποψή μου υπάρχει από ένα συγκεκριμένο κίνδυνο. Κίνδυνος διάβρωσης ε, του στρατιωτικού ε, δυναμικού των δυνατοτήτων που υπάρχουν στην Ευρώπη. Όσον αφορά τα στοιχεία για την άμυνα στην Ευρώπη, τα στοιχεία τα οποία έχει συγκεντρώσει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας καταδεικνύουν με απόλυτη σαφήνεια ότι εδώ και κάποια χρόνια οι δαπάνες ε, μειώνονται, συρρυκνώνονται σημαντικά. Γνωρίζουμε όλοι μας ε, πολύ καλά ότι η Ευρώπη διέρχεται μια δύσκολη οικονομική περίοδο είναι γενικώ απαραίτητο να μειωθούν οι ε, πόροι ε, και οι δημόσιες διαπάνες για να επανέλθει η σταθερότητα. Εγώ όμως παρόλα αυτά πιστεύω ότι ακριβώς επειδή υπάρχουν αυτές οι οικονομικές ε, δυσκολίες και από ό,τι φαίνεται δεν θα λυθούν σύντομα τα προβλήματα, είναι απαραίτητο να ληφθούν θραλές αποφάσεις στις δαπάνες για την άμυνα στο μέλλον κανένα από τα κράτη-μέλη δεν θα μπορέσει να θεωρεί ότι είναι ε, αυτάρκες ε, στον τομέα της άμυνας, ούτε σε επιχειρησιακό επίπεδο, ούτε σε επίπεδο πόρων ε, για την έρευνα, την ανάπτυξη, για την προσαρμογή των περίπλοκων συστημάτων εξοπλισμών. Αυτά που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια τα δείχνουν όλα αυτά με απόλυτη σαφήνεια. Λόγω του ότι έχουν περιοριστεί οι πόροι, σχεδόν όλα τα κρατημέλη μειώνουν τις δυνατότητές τους που πλέον είναι δαπανηρές στη συντήρηση. Όμως ε, με τέτοιου είδους επιλογές ε, το αποτέλεσμα είναι ότι η Ευρώπη στο σύνολό της χάνει, χάνει ακριβώς αυτές τις πολύ σημαντικές δυνατότητες που τις ε, δίνουν μια αυτονομία δράσης. Αν δει κανεί τα στοιχεία και για τις επενδύσεις στον τομέα της άμυνας, θα καταλάβει ποιο είναι το πρόβλημα. Ε, πάω πάλι στα στοιχεία της Υπηρεσίας Άμυνας της ΕΝΤΑ. Το 2010 τα 26 ε, κράτη συνολικά επένδυσαν 34 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση συστημάτων και εξοπλισμών και στρατιωτικών εξοπλισμών. Από αυτά τα 7,5 περίπου εκατομμύρια δόθηκαν σε προγράμματα, κοινά προγράμματα ε, που εφάρμοσαν πάνω από δύο κράτη-μέλη. Άρα δηλαδή μόνο το 22% των προγραμμάτων ευρωπαϊκών προμηθειών ε, επεκτάθηκαν σε περισσότερα από δύο κράτη-μέλη. Στην περίπτωση της έρευνας η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη. Περίπου 2 δισεκατομμύρια από τα 2,1 εκατομμύρια μόνο τα 246 εκατομμύρια, δηλαδή μόνο το 11,8% διοχετεύτηκε σε προγράμματα που εφαρμόστηκαν από δύο και περισσότερα κράτη-μέλη. Δηλαδή σήμερα στην Ευρώπη έχουμε μια πραγματικότητα όπου οι αποφάσεις που λαμβάνονται για την αγορά στρατιωτικών συστημάτων και ακόμα περισσότερο οι αποφάσεις για επενδύσεις στην έρευνα, οι αποφάσεις αυτές καθορίζονται από εθνικά συμφέροντα και αυτή είναι μια πραγματικότητα που δεν έχει καμία σχέση με τους πολιτικούς στόχους που είναι να γίνουν περισσότερα στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας και με τους οικονομικούς στόχους να τα καταφέρει κανείς, κανείς καλύτερα. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει σημαντική αύξηση της συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη-μέλη, έτσι ώστε από κοινού να αποφασίζουν πού θα κατευθύνουν τους πόρους τους και έτσι ώστε να υπάρχει μια ουσιαστική και καλή ε, στρατιωτική ικανότητα και δυνατότητες για το μέλλον. Να υπάρξει λοιπόν καταρχήν ε, πολιτική συμφωνία, δέσμευση των ε, κυβερνήσεων ε, και μεταξύ τους και απέναντι στην Ευρώπη. Αυτές λοιπόν οι αποφάσεις πρέπει να ενταχθούν μέσα στο οικονομικό πλαίσιο και στις οικονομικές σχολές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Βέβαια, μπορεί κανείς να προχωρήσει ευφυώς αναζητώντας την βέλτιστη δυνατή χρήση των δαπανών ε, με βάση την αρχή, τις αρχές της οικονομίας κλίμακας. Η ισορροπία στα δημόσια οικονομικά ε, νομίζω ότι είναι ε, η ισορροπία αυτή συμβαδίζει με την ανάπτυξη. Και γι' αυτό το λόγο Εάν συμβούν όλα αυτά, θα αυξηθεί και η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει ανταγωνιστικότητα και στον τομέα της ε, άμυνας. Ε, πρέπει να περιμένουμε περισσότερα από τους κοινού θεσμού και πρέπει να προσφέρουμε και περισσότερα. Μεγαλύτερη και καλύτερη συνεργασία για να προχωρήσει το ευρωπαϊκό σχέδιο. Είναι λοιπόν σαφές ότι μιλάμε για βήματα, για φάσεις. Το θέμα της κυριαρχίας των κρατών δεν είναι κάτι το δευτερεύον. Βέβαια, στον τομέα της άμυνας, ακριβώς όπως συνέβη και με το θέμα του νομίσματος, είναι απαραίτητο πρώτα απ' όλα να επιτύχουμε σύγκληση των εθνικών πολιτικών και κατόπιν να υπάρξει ουσιαστική ολοκλήρωση η οποία μακροπρόθεσμα θα σημαίνει και ε, υπερκέραση των εθνικών συμφερόντων. Είναι λοιπόν σημαντικό να υπάρξει επανεκκίνηση από ό,τι φαίνεται τώρα πια έχουμε την ευκαιρία της επανεκκίνησης γιατί με αρκετή οξυδέρκεια αποφασίστηκε το επόμενο Συμβούλιο του Κεμβρίου να ασχοληθεί με θέματα ευρωπαϊκής άμυνας. Θα ήταν αδύνατον να ολοκληρωθεί το Συμβούλιο οδηγώντας σε μείωση των ε, εισφορών για την άμυνα. Εγώ πιστεύω ότι εμείς οφείλουμε να επιτύχουμε δύο βασικούς στόχους. Ο πρώτος είναι να επαναβεβαιώσουμε με απόλυτη σαφήνεια ότι η άμυνα είναι σημαντική και ότι η άμυνα δεν είναι απλά έκφραση ισχύω. Αντίθετα, είναι έκφραση αποφασιστικότητας για να υπαγορεύσει κανείς τους όρους για την ειρήνη και την ανάπτυξη. Ο δεύτερος ε, στόχος είναι το να υπάρξει ε, μια νέα φάση προγραμμάτων και σταδιακών βημάτων. Στο επόμενο Συμβούλιο, το σημείο κίνησης για να προχωρήσουμε γρήγορα είναι να υπάρχει μεγαλύτερη ολοκλήρωση και καλύτερη συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Η άμυνα δεν μπορεί να περιθωριοποιηθεί στο πλαίσιο των αποφάσεων που καλούνται να λάβουν ε, οι κυβερνήσεις κατά τα επόμενα έτη. Η άμυνα είναι καθοριστική σημασίας γιατί είναι διατομεακή και διότι ε, προϋπάρχει σε οποιαδήποτε πολιτική επιθυμεί κανείς να εφαρμόσει. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε όλα αυτά που σας λέω καλύτερα βλέποντας ε, και την προσφορά της Ιταλίας στο Αφγανιστάν. Η Ιταλία έχει προσφέρει πάρα πολλά και έχει προσφέρει τόσο σε επίπεδο δαπανών όσο και σε επίπεδο διεθνούς συνεργασίας. Η άμυνα λοιπόν είναι καθοριστική σημασίας για να διασφαλίζονται τα συμφέροντα της Ευρώπης και είναι καθοριστική σημασία για να υπάρχει και ισορροπημένη σχέση με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Αυτό είναι προϋπόθεση για να επανακαθορίσουμε τη σχέση μας ε, με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Η άμυνα είναι καθοριστική σημασία και για επενδύσεις στην άμυνα κυρίως ε, σε τομείς ε, τεχνολογία εχμή. Άρα δηλαδή πρέπει να ληφθούν οι σωστέ αποφάσει σε επίπεδο Ευρώπης και η Ιταλία προτίθεται να συνδράμει έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη διαχείριση της κρίσης. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι είναι απαραίτητο να υπάρξουν οικονομικές θυσίες ε, και επίσης ε, γνωρίζουμε ή έχουμε συνειδητοποιήσει τις ευθύνες μας. Είμαστε αποφασισμένοι να τιμήσουμε τις ε, ευθύνες μας ακόμα και κατά τη διάρκεια της Ιταλικής Προεδρίας έτσι ώστε να προχωρήσει η Ευρώπη ως ένας καθοριστικός παράγων ο οποίος θα είναι και σε θέση να διαδραματίσει το ρόλο στον οποίο προσβλέπουμε όλοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και βεβαίως είμαι στη ε, διάθεσή σας ε, για να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ. Μάριο, βλέπω ότι έχεις κάνει ήδη μια καλή αρχή στα νέα σου καθήκοντα και συμβάλλεις σε αυτά που συζητήσαμε μετά από την παρουσία του κυρίου Γενικού Γραμματέα σε ό,τι αφορά τις εργασίες της Επιτροπής και της Επιτροπής μας στα πλαίσια της άμυνας, αλλά και σε ό,τι αφορά και άλλα επίπεδα προετοιμασίας της Συνόδου του Δεκεμβρίου θα είναι μια σύνοδος όπου θα τεθούν και θα πρέπει να τεθούν οι απαραίτητοι στόχοι και οι τρόποι επίτευξής τους. Πολλά από τα πράγματα τα οποία θεωρούμε αυτονόητα δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμα, περιλαμβάνονται στη συνθήκη της Λισαβόνας σε ό,τι αφορά τα, τις, ομάδες, ε, τις μάχημες ομάδες, για παράδειγμα, οι οποίες έχουν οριστεί στη θεωρία, αλλά δεν έχουν εφαρμοστεί όλα αυτά στην πράξη. Επίσης, σε ό,τι αφορά την θεσμοποιημένη μόνιμη συνεργασία, ένα από τα βασικά εργαλεία, προκειμένου να σημειωθεί πρόοδος για όσους το επιθυμούν. Δεδομένης της ομοφωνίας που ε, επικρατεί ως προϋπόθεση, θεωρώ ότι το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό σε ό,τι αφορά δηλαδή όσους θέλουν να προχωρήσουν περαιπέρα και σε όσους ούτε επιθυμούν για διάφορους λόγους. Όλα αυτά θεωρώ ότι θα πρέπει να πάρουν τη σειρά τους μετά τη συνθήκη της Λισαβόνα που θα έχει κλείσει τρία χρόνια κατά τη χρονική συγκυρία της ε, Διεξάγωγή τη ε, διάσκεψη κορυφή. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να κινηθούμε προ την κατεύθυνση αυτή του επόμενου μήνε. Ο κύριος Τανζάν και ο κύριος Σαλαφράγκα. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, αγαπητέ Μάριο, ως ευπαρέστης ε, η Υποεπιτροπή Άμυνας ε, και Ασφάλειας είναι ιδιαίτερα ευτυχής για αυτό το διορισμό και πιστεύω ότι θα είναι πολύ ε, σημαντική αυτή η διαφορά, γιατί θα ξέρουμε, αν μη τι άλλο, τις εκθέσεις μας θα τις διαβάζει ένας ε, υπουργός άμυνας, ε, που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος στις απόψεις και την ευήκον στις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε ό,τι αφορά το Συμβούλιο για τα τέλη Δεκεμβρίου, έχω δύο σχόλια και μία ερώτηση. Όπως ακούσαμε και στην ομιλία, το πιο σημαντικό θέμα είναι η ανάγκη να πάμε ακόμη πιο μακριά από κοινού. Γιατί είναι τέτοια η δημοσιονομική λιτότητα που κανένα κράτο μέλος από μόνος του δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στις ε, στρατιωτικέ ε, προκλήσεις και τις προκλήσεις στρατιωτική ικανότητα των μέλλον. Οπότε, βέβαια θα πρέπει να στηριχθούμε και στις μεμονωμένες ε, ικανότητε των κρατών μέλων. Αλλά δούμε το χάρτη, ε, βλέπουμε ότι μόνο δύο χώρε συμβάλλουν πάνω από το 50% των ευρωπαϊκών ικανότητων. Η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο ε, βλέπουμε ότι ε, συμβάλλει περισσότερες σε αμυντικές προσπάθειες. Οπότε πώς θα παροτρύνουμε και τα υπόλοιπα κρατημέλη να καταβάλουν τις απαραίτητες προσπάθειες και μεμονωμένα ώστε η συλλογική προσπάθεια είναι ακόμη πιο ενισχυμένη. Δεύτερο θέμα αφορά τις, ε, την πολεμική βιομηχανία που ξέρουμε ότι στην Ευρώπη η αμυντική βιομηχανία είναι πολύ παραγωγική αλλά θα μπορούσε να γίνει ακόμη πιο ανταγωνιστική με αναδιαρθρώσεις, με αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Η Επίτροπη Ταγιάννη και Μπαρνιέ θα υποβάλουν σχετικές προτάσεις και στο δημοσιονομικό πλαίσιο και τις, το πλαίσιο της λιτότητας που ταλανίζει όλα τα κράτη-μέλη, ξέρουμε ότι οι αναδιαρθρώσεις μπορούν να οδηγήσουν σε απόλυτη θέση αναπασχόληση, σε κλείσιμο μερικών βιομηχανιών και κανένα κράτος μέλος δεν είναι έτοιμο να ανλάβει αυτό το τίμημα βραχυπρόθεσμα. Και μάλιστα η Ιταλία έχει πολύ ε, αποδοτική πολεμική βιομηχανία, αμυντική βιομηχανία, ε, πώς ε, γίνεται στην Ιταλία αυτή η συζήτηση για την αναδιάρθρωση αμυντικής βιομηχανίας και τρίτον για τις προτεραιότητες του Συμβουλίου Άμυνας που θα αφιερωθεί στη, σε θέματα άμυνας. Ενίσχυση της ικανότητας. Όπως είπε και πριν από λίγο ο Γενικός Γραμματέας, τι μας ε, ενδιαφέρουν οι ικανότητες, αν δηλαδή δεν υπάρχει βούληση για τη χρησιμοποίησή τους. Και αυτό που ίσως λείπει είναι ακριβώς η πολιτική θέληση στο μέλλον ε, ε, διαπιστωθεί έλλειψη αυτή η πολιτική βούληση για δράση. Και ε, το θέμα είναι ποιες προτεραιότητες θα πρέπει να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση να τις καθορίσει πρώτα σε θέματα εξωτερικής πολιτικής πριν ξεκινήσει μια αμυντική πολιτική και το συζητήσαμε αυτό το θέμα μακρόν στην Υποεπιτροπή Ασφάλεια και Άμυνα. Μια μεθοδολογία όπω η Λευκή Βίβλος που έγινε στη Γαλλία, μια τέτοια Λευκή Βίβλος σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωσης, δηλαδή δεν θα ήταν ένα κατάλληλο διάβημα για να κάνουμε τουλάχιστον μια παρήθμιση των προτεραιοτήτων μα που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για θέματα άμυνα. Ευχαριστώ. Ο κύριο Αλαφράγκα, ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να πω ότι όταν ε, είδα το σημείο 5 στην ημερήσια διάταξη, ανταλλαγή απόψεων με τον Μάριο Μάωρο, Υπουργό Άμυνας της Ιταλίας, αισθάνθηκα μια μεγάλη προσωπική ικανοποίηση. Γι' αυτό και θα ήθελα, αγαπητέ Μάριο, αγαπητέ Υπουργέ, να σας συγχαρώ θερμά για το διορισμό σου. Και θα ήθελα ε, και προσωπικά, αλλά και εκ μέρους ομάδας, να σας διαβάσω θερμές ευχές για καλή επιτυχία στην ε, διεξαγωγή των καθηκόντων σου και ήταν πολύ χρήσιμη αυτή η ευκαιρία που έχουμε. Θα ήθελα να υποβάλω δύο ερωτήσεις. Σίγουρα ο υπουργό ε, ε, έδειξε ιδιαίτερη ε, ευαισθησία και επένδυση στο Κοινοβούλιο, αλλά και στις επισκέψεις των επιχειρήσεων στην ΙΣΑΦ. Ποια είναι η γνώμη της Ιταλίας για το τι θα γίνει μετά το 2014, γιατί οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, θέλουν να διαπραγματευτούν ένα σύμφωνο ασυλίας για τα στρατεύματα. Η Γερμανία θα περιορίσει ε, τις δικές αποστολές, οπότε τι θα γίνει με τις νέες υποχρεώσεις που θα έχει η διεθνής κοινότητα για ε, αξιολόγηση, παροχή συμβουλών, ε, κατάρτιση. Ποια είναι η θέση σας γι' αυτό. Επίση, πέραν των πολύ εύστοχων ερωτήσεων του συναδέλφου Ντανζάν για την πολιτική ασφάλεια και άμυνα, θα ήθελα να συζητήσουμε με τον αγαπητό πρώην συνάδελφο Μάριο Μαώρο πώς βλέπει την κατάσταση στη Συρία. Ο Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ ζήτησε από τα μέλη του ΝΑΤΟ ε, να προβλέψουν κάποια σχέδια δράση ε, σε περίπτωση επίθεση με χημικά όπλα. Το περασμένο Σάββατο είδαμε τι έγινε. Υπάρχει ένα κίνδυνο να πυρποληθεί ολόκληρη η περιοχή. Επίση ακούσαμε δηλώσει ε, των ε, Υπουργών τη Γαλλία και του Ηνωμένου Βασιλείου. Και ο Γενικό Γραμματέας του ΝΑΤΟ είπε ότι η πιο κατάλληλη είναι μια πολιτική λύση τέθηκε και η πρόταση για μια ζώνη αποκλεισμού των πτήσεων, αντίστοιχη με αυτή που εφαρμόστηκε στη Λιβύη. Η Ιταλία τι γνώμη έχει για την κατάσταση αυτή την τραγική κατάσταση στη Συρία και ποια θα ήταν η καλύτερη διέξοδος εν ώψη της απόφασης του Ιουνίου όπου θα συζητηθεί και το θέμα του εμπάργου από τους Ευρωπαίους Υπουργούς. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Μάριο Μάριο, κύριε Υπουργέ, λυπάμαι, σας αποκαλώ ακόμα Μάριο. Συγχαρητήρια για τον διορισμό μας. Θα θέσω κάποια από τα ίδια ερωτήματα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα Αφγανιστάν μετά το ΕΖΑΦ. Είσαστε πεπισμένος ότι υπάρχουν αρκετές δυνάμεις που έχουν μείνει πίσω σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση για να διασφαλίσουν ότι τα λιμπάν δεν θα ξαναπάρουν το πάνω χέρι. Ιδάλλως θα θεωρηθεί τεράστια σπατάλη χρημάτων και ενέργειας και δυναμικού και προσωπικού και ενόπλων δυνάμεων, αν επανέλθουμε στην προηγούμενη κατάσταση. Και τι θα κάνει η Ιταλική κυβέρνηση προκειμένου του Αφγανιστάν να παραμείνει ελεύθερο από τους Ταλιμπάν στο μέλλον για να έχει νόημα και η αρχική επιχείρηση σε ό,τι αφορά επίσης ξέρω ότι στην προηγούμενη ιδιότητά σας ως μέλος της Επιτροπής σας ενδιαφέραν πάρα πολύ οι χριστιανοί στην Συρία, για παράδειγμα, που αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα, τεράστιους κινδύνους σε περίπτωση που θα ε, επικρατήσουν οι σολαφιστές. Το Ισραήλ έχει επέμβει κατά μεταφοράς όπλων από τη Χεσβολά από την κυβέρνηση του Ασάντ. Φαντάζομαι ότι υπάρχει πραγματικό ενδεχόμενο να ξεσπάσει πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Συρία και να υπάρξει και εμπλοκή του Ιράν. Δεν ξέρω αν θεωρείτε ότι ανησυχώ υπερβολικά. Πείτε μου ποιε είναι οι δικές σας σκέψεις. Αν υπήρχε τέτοια πρόθεση να επέμβουμε, θα ήταν όπως το Μάλι ένα ε, συνασπισμός, μια συμμαχία όσων θέλουν να προχωρήσουν. Τι μορφή θα έπαιρνε με τέτοια παρέμβαση και τέλο ότι αφορά την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία άμυνας. Η ομάδα μας είναι αρκετά σκεπτικιστική σε ό,τι αφορά αυτά που έχουν επιτευχθεί ως τώρα. Ένα από τα θέματα είναι και ο ενέργειος ανεφοδιασμός. Τι πιθανότητε έχει η υπηρεσία να προσφέρει κάτι, να πετύχει μεγαλύτερη δυνατότητα, μεγαλύτερη ανάπτυξη δυναμικού pooling and sharing προκειμένου να δικαιολογήσουν την ε, ανάγκη ύπαρξης ε, του EDA με 26 κρατημέλη στην παρούσα φάση, εκτός από την Δανία δηλαδή, όλοι εκτός από την Δανία. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ, ο κύριος να σας ε, συγχαρώ και εγώ. Αναφερθήκατε στην διάσκεψη κορυφής του Δεκεμβρίου που έχει αφιερωθεί στην Ευρωπαϊκή Άμυνα. Θα ήθελα λοιπόν και εγώ να υπογραμμίσω τρία-τέσσερα ζητήματα σχετικά με την ε, διάσκεψη αυτή. Η ΚΕΠΑ θεωρώ ότι ως εργαλείο θα μπορούσε να μας προσφέρει πολύ περισσότερες ευκαιρίες για ανάληψη δράσης από ό,τι μας προσφέρει στο παρόν. Και τονίζω ιδιαίτερα το σκέλος της ανάπτυξης ικανοτήτων για την διεξαγωγή των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και για να αντιμετωπίσουμε την έλλειψη ε, συντονισμού. Πρώτη λοιπόν παρατήρηση. Το κέντρο επιχειρήσεων που ατέθηκε σε δράση στις αρχές του περασμένου έτους αποτελεί μία βάση για τις μόνιμες αστυνομικέ δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι υπεύθυνο για την ε, προγραμματισμό των τρέχουσών και των μελλοντικών επιχειρήσεων. Εγώ θεωρώ ότι είναι ένα βήμα προς την διαμόρφωση ενός αρχηγείου ευρωπαϊκού, αν θέλετε, μελλοντικά. Ποια είναι η δική σας άποψη και θα ήθελα να σας καλέσω προς αυτή την κατεύθυνση να κινηθείτε. Κατά δεύτερον, συζητούμε ακόμα το ρόλο και την έννοια των ε, μάχημων ομάδων. Ως πρώην υπουργό Άμυνα θυμάμαι διάφορες συζητήσεις ε, επ' αυτού σε Ευρωπαϊκά Συμβούλια. Οι συζητήσεις αυτές έμεναν πάντοτε ατελώς φορές σε ό,τι αφορά ενδεχόμενο ρόλο των μάχημων ομάδων, σε ό,τι αφορά την ε, αρχική τους δράση ή την χρήση του ως ομάδες επιχειρησιακής ε, συμπληρωματικότητας. Ίσως θα μπορούσατε να τονίσετε ποιο είναι ο ρόλος τους στα πλαίσια της επιστολής της Βαϊμάρης που υπογράφηκε το 2010 και των σχετικών προτάσεων που έγιναν πιο πρόσφατα και τέλος ποια είναι η άποψή σας σε ό,τι αφορά τη χρήση των θεσμών και των διαδικασιών που εισήχθησαν με τη συνθήκη της Λισαβόνας και που έχουμε στη διάθεσή μας. Για παράδειγμα, η μόνιμη διαστρωμένη συνεργασία. Η πρωτοβουλία ανάπτυξης δυναμικού που ονομάζεται Pooling and Sharing. Σας παρατρύνω λοιπόν και πάλι προς την κατεύθυνση αυτή να κινηθείτε. Ευχαριστώ, κύριε Γιαννάκου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ τον συνάδελφο κύριο Μάουρο ε, όχι μόνο για την ε, θέση την οποία κατέλαβε, αλλά και για όσα είπε προηγουμένως σχετικά με την Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ασφάλεια. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ε, το κόστος στην Ευρώπη είναι πολύ μεγαλύτερο για πολύ λιγότερη αποτελεσματικότητα. Όλοι το γνωρίζουμε αυτό. Έχει υποθεί από την πρώτη στιγμή το 2001 όταν άρχισαν οι συζητήσεις για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Άμυνας και Ασφάλειας αλλά βέβαια η υπόθεση της ομοφωνίας δημιουργεί συγκεκριμένα προβλήματα στο να προχωρήσουν τα ζητήματα αυτά. Και ίσως ο μοναδικός τρόπος θα ήταν η ενισχυμένη συνεργασία, κύριε Υπουργέ, διότι είναι γνωστό ποιοι έχουν σοβαρές αντιρρήσεις για, το, για την πρόθεση όσων είπατε προηγουμένως. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί και να ξεπεραστεί. Ε, οι χώρες μας είναι μέλη του ΝΑΤΟ, οι περισσότερες. Αυτό δεν σημαίνει ότι παρακάμπτουμε το ΝΑΤΟ ή ότι δεν θέλουμε την ύπαρξή του, αλλά είναι ανάγκη να γίνει ένα συνεκτικό σύστημα αντιμετώπισης των προβλημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία άλλωστε ξοδεύει πάρα πολλά, όπως είπατε, σε βοήθεια, διοικητική υποστήριξη, ανάπτυξη κλπ. Πολύ περισσότερα από όσα διαθέτουν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Επομένω, το Συμβούλιο του Δεκεμβρίου νομίζω ότι πρέπει να αναμένουμε μια τελείως διαφορετική προσέγγιση του θέματος και ίσως εσείς θα μπορούσατε να μας πείτε ποιες θα ήταν οι δύο-τρεις προτάσεις συγκεκριμένες που η Ιταλία θα επεδίωκε και στα ζητήματα που αναφέρατε και, στα, ε, και στη συνεργασία και στην κατάρτιση και εκπαίδευση. Παραδείγματο χάρη τι γίνεται με το σύστημα το οποίο είχε αποφασιστεί και το οποίο υπονομεύεται εσωτερικά για την κατάρτιση και εκπαίδευση και τη συνεργασία στελεχών των στρατιωτικών δυνάμεων της Ένωσης. President, Paramount President Ο πρώην πρόεδρος Pöttering, ευχαριστώ πολύ πρόεδρε και σας καλωσορίζω και σα συγχαίρω κύριε Υπουργέ Μάιρο Μάρο. Είναι θαυμάσιο το ότι σε βλέπω εδώ σήμερα ω Υπουργό Άμυνα τη Ιταλία, Πάντα πίστευα στην Ιταλία και το γεγονό ότι σε διόρισαν Υπουργό ε, Άμυνα δικαιολογεί την πίστη μου στην Ιταλία. Αν μου επιτρέψει να σου μιλάω στον ελληνικό, μίλησες για ένα όραμα. Και ο Αλτσίδε Γκάσπερη και ο Κόντον Άντενάουερ εξέφρασαν το όραμα της δεκαετίας του 50 για τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης Άμυνας με έναν Ευρωπαϊκό στρατό. Και νομίζω ότι χρειαζόμαστε και πάλι στόχους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει τον ε, όρο Ευρωπαϊκό Στρατό να το χρησιμοποιούμε και πάλι, γιατί μας δίνει μια ορισμένη κατεύθυνση και μιλήσατε και για τις ε, μάχημες ε, ομάδες, τις ομάδες μάχης. Θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα πυρήνα για ένα Ευρωπαϊκό Στρατό. Και ακούω από πίσω μου τους βρετανού συναδέλφους να στενάζουν. Δεν χρειάζεται να συμμετέχουν, άμα δεν θέλουν να συμμετέχουν. Μπορεί να είναι μια διατρομένη συνεργασία, αλλά εγώ θα ήθελα να εισαγάγουμε εκ νέου έναν ε, τέτοιο στόχο και ένα όρο με όραμα για την ευρωπαϊκή συνεργασία. Σου εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο σου, αλλά και σε σένα και σε όλη την Ιταλική κυβέρνηση. Thank you, Herr President. Now, Mr. Van Orden. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Van Orden. Uh, um, Ευχαριστώ και συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια κύριε Υπουργέ, για το διορισμό, για το διορισμό σας. Και ευχαριστώ για την επιβεβαίωση που μας κάνετε για το τι σημαίνει η ΚΕΠΑ. Διεύρυνση της ε, Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Αυτό είναι ο πρωταρχικός στόχος της ΚΕΠΑ και ήταν ε, σαφέστατα και από τα δικά σας λεγόμενα και σας ευχαριστώ για αυτή την ενάργεια και τη σαφήνειά σας. Έχω δύο ερωτήσεις. Τι ε, βήματα θα πραγματοποιήσει η Ιταλία για να μπορεί να αναπτύσσει περισσότερες στρατιωτικές δυνάμεις να μπορεί να αυξήσει τη δυνατότητα ανάπτυξης. Θέλετε να ενισχυθεί και το ΝΑΤΟ. Ποια είναι η γνώμη της Τελεία σχετικά. Η ε, κυρία Μαρτίνη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ, αγαπητέ Μάριο. Θέλω να εκφράσω και δημόσια τη χαρά μου για το διορισμό σου. Ε, εγώ μπόρεσα να έρθω εδώ και λόγω της δικής μου της απόφασης ε, να μην εκλεγείς στην ε, ε, Βουλή, στην Γερουσία της Ιταλίας. Τώρα λοιπόν, με τη δική δικό στο διορισμό, πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ γιατί η Ιταλία δείχνει ότι είναι περισσότερο ευρωπαϊκός προσανατολισμένη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Αγκουράκης. Κύριε Αγκουράκη, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, ε, καταρχήν θα ήθελα να ρωτήσω τον, τον Υπουργό αν θεωρεί την πρόσφατη επίθεση του Ισραήλ στη Συρία ως μια πράξη εισβολής και παραβίασης εδαφικής ακεραιότητας μιας χώρας από μια άλλη χώρα. Το δεύτερο ζήτημα που ήθελα να το ρωτήσω είναι το εξή. Όντως γίνεται αυτή η συζήτηση και το τελευταίο καιρό και γενικότερα για τις διάφορες μορφές αμυντικής συνεργασίας μεταξύ χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Battle groups, ο συνάδελφος από την Πολωνία αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία της Βαϊμάρης, υπάρχει συνεργασία Γαλλίας με Ηνωμένο Βασίλειο κτλ. Ε, ποια είναι η γνώμη του Υπουργού. Γιατί, γιατί δεν προχωράνε, εγώ λέω ευτυχώ που δεν προχωράνε, χαίρομαι για αυτό το λόγο και έχω και μια εξήγηση η ο λόγος που αυτές οι συνεργασίες δεν προχωράνε και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι επειδή οι χώρες ντρέπονται να χρησιμοποιήσουν τη την στρατηγική ισχύ για στόχους που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και γι' αυτό θέλουν την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε ενωμένε να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα. Παράδειγμα Μαλή. Γιατί, γιατί με τη Γαλλία δεν πήγε κανένα άλλος στο Μάλι. Θα μπορούσαν να πάνε. Δεν πάνε. Και αλλού υπάρχουν τέτοιες ε, δυνατότητες. Και εγώ νομίζω δεν γίνεται αυτό το πράγμα ακριβώ γιατί οι, οι, λόγοι που υπάρχουν τέτοιες επεμβάσεις είναι αντίθετες με το διεθνές δίκαιο. Τέλος, επειδή έγινε λόγος για την αμυντική βιομηχανία, κύριε Υπουργέ, και όχι πρώτη φορά, έγινε και τώρα. Και επειδή και εσείς χρησιμοποίησατε τον όρο ανταγωνιστικότητα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό στην πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα σημαίνει να εξαφανιστούν υπόθηκε κιόλα από κάποιον από τους συνομιλητές μας, ένα μεγάλο μέρος από τις αμυντικές βιομηχανίες Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως έγινε και με ένα μεγάλο αριθμό βιομηχανιών ως συνέπεια της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς. Αυτό θέλουμε. Ανταγωνιστική αμυντική βιομηχανία σημαίνει παραδείγματο χάρη οι 2.000 εργαζόμενοι των ελληνικών αμυντικών συστημάτων σήμερα στην Ελλάδα, οι οποίοι είναι απλήρωτοι για ένα χρόνο, τελειώνω Πρόεδρε, να, χάσουν εντελώ τι δουλειέ του. Πώ θα λυθούν αυτά τα προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ. Grazie. Πριν λοιπόν ε, δώσω το λόγο στον Υπουργό για τις απαντήσεις του, θα ήθελα και εγώ να σας ε, συγχαρώ γιατί πραγματικά Είσαστε ανεκτήμητος για τη χώρα μας. Και επιτρέψτε μου να κάνω κι εγώ μία παρατήρηση και να υποβάλω και μία ερώτηση. Αναφέρομαι στο πρώτο κομμάτι της ε, παρέμβασής σας. Νομίζω ότι είναι δύσκολο να προχωρήσουμε προς ουσιαστική βελτίωση στον τομέα της ε, άμυνας και στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι δύσκολο διότι αυτές οι δύο ε, πολιτικές σε τελική ανάλυση είναι τα προπύργια της εδαφικής κεραιότητας του κάθε κράτους που καλείται να εκχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά θα μπορούσαν να συμβούν μόνο εφόσον σημειωθεί και ουσιαστική πολιτική και θεσμική πρόοδος. Κατόπιν τούτου, όποιος βέβαια είναι πεπισμένος για όλα αυτά, πιστεύει ότι πρέπει καταρχήν, όπως είπα, να υπάρξει πολιτική ολοκλήρωση. Μία ερώτηση τώρα. Ε, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ζητούν από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμβάλλουν περισσότερο στην ε, πολιτική άμυνας. Υπάρχει αυτό το αίτημα αφενός των ΗΠΑ, αφετέρου υπάρχουν οι Υπάρχει κρίση οικονομική, δημοσιονομική που πλήττει πολλά κράτη και την Ιταλία. Κύριε Υπουργέ, εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει ένα περιθώριο ε, εξοικονόμησης δαπανών μέσα, παραδείγματος χάρη από την απλούστευση των εξοπλιστικών συστημάτων και αν θέλετε και μέσα από τη βελτίωση πολιτικών εξοπλισμού των μεμονωμένων κρατών μελών. Δηλαδή υπάρχει εκεί κάποιο περιθώριο να προκύψουν εξοικονομήσεις ε, πόρων και κοντιλίων. Ευχαριστώ πολύ. Όπως σας είπα και κατά τη διάρκεια της παρέμβασής μου, εγώ ε, ήθελα να ξεκινήσω τη ανάληψη καθηκόντων επισκεπτόμενος τα στρατεύματα στο Αφγανιστάν. Εχθές συναντήθηκα με το γενικό ε, με τον ε, επικεφαλής των δυνάμεων Άισεφ και τον πρόεδρο Καρτσάη στο Αφγανιστάν. Γι' αυτό λοιπόν θα απαντήσω καταρχήν στις ερωτήσεις μου ετέθησαν για τη στρατηγική μετά το 2014, κυρίως όσον αφορά στο Αφγανιστάν. Η θέση Ιταλίας είναι ξεκάθαρη. Εμείς δεν προτιθέμεθα επουδενή να ξεχάσουμε όλα αυτά που επιτεύχθηκαν ώστε να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος στο Αφγανιστάν. Επισκέφθηκα τη ώρα το Φαράτα, το συντάτη τις βάσεις μας εκεί, όπου έχουν αναπτυχθεί οι περίπου 4.000 άνδρες Ιταλοί. Και στις συζητήσεις που είχαμε τον στρατηγό Ντάμφορτ, τον επικεφαλής ε, του, της ΙΣΑΦ, ξεκαθάρισα ότι μετά το 2014 θα πρέπει να ισχύσει η αρχή της αναλογικότητας και με βάση όλα αυτά που έχουν επιτύχει τα κράτη της ΆΙΣΑ. Άρα δηλαδή η Ιταλία μετά το 2014 αναλογικά πάλι θα συμμετάσχει για να διασφαλίσει την παρουσία ανδρών, την οικονομική συνεργασία τόσο όσον αφορά την υποδομή, την εκπαίδευση, τα θέματα υγείας, ε, την προάσπιση και την προαγωγή της των δύο φύλων, όσο και πάρα πολλά άλλα. Εν πάση τόση όλα αυτά που στο Αφγανιστάν επιτεύχθηκαν χάρη της παρουσίας των στρατιωτικών δυνάμεων που ε, διασφάλισαν αυτή την πρόοδο. Έτσι λοιπόν, όπου δεν υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες, Σημαίνει αυτό σε κάποιες περιοχές. Εκεί υπάρχει λιγότερη πρόοδο στο Αφγανιστάν. Όλα αυτά τα είπα και στον πρόεδρο Καρζάη. Και επίσης του εξήγησα με λεπτομέρειες της ε, συμφωνίας τις συμφωνίες που έχουν επιτευχθεί, γιατί η συμμαχία δεν είναι μόνο στρατιωτική, είναι και πολιτικής φύσεως. Άρα δηλαδή μιλάμε για ξεχωριστές συμφωνίες που έχουν συναυτεί με τις αρχές του Αφγανιστάν για να υπάρχει ασυλία για τους στρατιώτες που βρίσκονται εκεί. Έχουμε λάβει σαφέστατη οντελή από διεθνείς ε, οργανισμούς. Αυτό σημαίνει όπου δραστηριοποιούμεθα, όπως και στο Λίβανο. Και όλα αυτά γιατί έχουμε ένα κοινό όραμα. Φτάνω λοιπόν στο διατάφτα. Είναι αλήθεια ότι ξεκίνησα τη θητεία μου, ανέλαβα ε, το αξιωμά μου ξεκινώντας ε, από το Αφγανιστάν αλλά πρέπει να σας πω φοβόμουν πιο πολύ τις ερωτήσεις που θα μου κάνατε εσείς από ό,τι όταν πήγα στο Αφγανιστάν κυρίως τις ερωτήσεις των ε, Ντανζόν και Βανόρντεν. γι' αυτό λοιπόν επιτρέψτε μου να εστιάσω την προσοχή μου σε κάποιες από τις ερωτήσεις τους γιατί οι ερωτήσεις που έκαναν καταδεικνύουν με απόλυτη σαφήνεια ότι πράγματι ε, μπορεί να υπάρξει ένα κοινό όραμα αν ο καθένας ε, κάνει σωστά τη δουλειά του. Και θα ε, αναφέρω το τι έκανε ας πούμε ο κύριος Μόντις αυτό το 1,5 χρόνο που είχε την κυβέρνηση η Ιταλία δεν ζήτησε ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Σταθερότητας. Η Ιταλία τα κατάφερε με τις δικές της δυνάμεις να λύσει τα προβλήματά της και να αντιμετωπίσει τα χρέη της. Και όχι μόνο αυτό, αλλά η Ιταλία ήταν στην πρώτη γραμμή για να στηρίξει χώρες όπως η Ελλάδα και επίσης και σε στρατιωτικό επίπεδο η Ιταλία και στο παρελθόν αλλά και στο μέλλον με επιμονή θα υπεραμεινθεί της άμυνας, όχι όμως ως έκφραση ισχύου, αλλά της άμυνας ως μια απαραίτητη προϋπόθεση για να διασφαλίσει κανείς την ειρήνη και την ανάπτυξη των λαών. Έτσι λοιπόν η συζήτηση που έχει ξεκινήσει στο Κοινοβούλιο μας για θέματα προϋπολογισμού και αμυντικών δαπανών, η συζήτηση είναι αυτή ε, θα περιλάβει ε, και βεβαίως στοιχεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Γιατί πιστεύουμε ότι μέσα από την κοινή άμυνα μπορούμε να λάβουμε καλύτερα και τις ευθύνες μας ε, ως κράτη. Θέλω να κάνω προβώ και σε άλλες διευκρινήσεις. Πολλοί συνάδελφοι ενθάρρονται απογοητευμένοι, επιφυλακτικοί Θέλω λοιπόν να πω ότι όποιος είναι ευρωσκεπτικιστής δεν είναι ότι βασίζεται μόνο σε κάποια επιχειρήματα, αλλά αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι δεν είναι πεπισμένος, δεν πιστεύει στην Ευρώπη. Εγώ λοιπόν δεν νομίζω ότι στο Συμβούλιο του Δεκεμβρίου μπορούμε να πάμε πιστεύοντας ακόμα ότι μπορούμε να ε, διαπραγματευόμεθα ή να αμφισβητούμε τα περιφερειακά θέματα όπως για κάποιους είναι οι μάχημες ομάδες, τα battle groups. Εκείνο που πρέπει να υπάρξει είναι να μπορέσουμε να κατανοήσουμε ότι η Ευρώπη θα ολοκληρωθεί μόνο με μια ευρωπαϊκή μέθοδο. Και η μέθοδος αυτή δεν είναι ε, μια μέθοδο που ξεκινάει από τη θεωρία και πάει στην πράξη, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Πάντα υπήρχε μια ρεαλιστική βάση, παραδείγματο χάρη, στην κοινή αγορά. Ξεκινήσαμε από τον άνθρακα και το χάλιβα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από την άμυνα. Αυτή είναι μια απαραίτητη προπόθεση για να μπορέσουμε να επιτύχουμε το όραμά μα. Και μάλιστα να διατηρήσουμε την ρεαλιστική μα αυτή στάση. Και θα αναφέρω συγκεκριμένο παράδειγμα. Στην Ιταλία πολλοί διαφωνούν για τα συστήματα άμυνας που πρέπει να υιοθετήσει ε, το Ιταλικό, να αγοράσει ε, το Ιταλικό κράτος. Μερικοί είναι υπέρ των F-35, άλλοι προτιμούν άλλα ε, συστήματα. Τώρα, αν περιοριστούμε στο είδος των αεροσκαφών και όχι στο ευρύτερο όραμα, καταλαβαίνετε ότι δεν θα κατανοήσουμε ότι μόνο μία ολοκληρωμένη άμυνα μπορεί να είναι αποτελεσματική. Το γεγονός λοιπόν ότι πρέπει να προβούμε σε ορισμένες συγκεκριμένες επιλογές, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να συμβαδίζουν επιλογές μας με τις επιλογές των ε, συμμάχων. Και αυτό πάλι δεν σημαίνει ότι ε, γίνεται για να υπεραμεινθούμε της ευρωπαϊκής ε, αμυντικής πολιτικής, αλλά διότι θέλουμε να υπεραμεινθούμε του οράματός μας. Αυτό που είπε ο κ. Βανόντεν σχετικά με το μέλλον του ΝΑΤΟ. Το πώς μπορεί κανείς να ενισχύσει το ΝΑΤΟ. Θέλω να πω το εξής. Τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ε, στην πλειοψηφία τους μέλη του ΝΑΤΟ. Άρα δηλαδή μια πιο δυνατή Ευρώπη, ε, πιο ολοκληρωμένη στρατιωτικά θα ενισχύσει το ΝΑΤΟ. Γι' αυτό λοιπόν εγώ πιστεύω ότι ακόμα και από το πρίσμα της ε, Μεγάλης Βρετανίας και όταν μιλάω για Μεγάλη Βρετανία μιλάω περισσότερο για μια κουλτούρα η οποία έχει άλλοι τους δεσμούς φυσικούς δεσμούς, αν θέλετε, με, την, ε, ε, με τον ευρωπαϊκό ε, τρόπο ζωής. Ας μην το ξεχνάμε αυτό. Ο, ε, στρατηγός Βαν Όρντεν θα θυμάται κάτι που είπε ο Τσόρτσιλ κατά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο στη μάχη της Αγγλίας και είπε ότι ποτέ τόσοι πολλοί δεν όφυλαν τόσα πολλά σε τόσο λίγους. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι εάν οι 750 ευρωβουλευτές μαζί με τους υπουργούς, αν όλοι αυτοί έχουν ένα κοινό όραμα, ποτέ τόσοι πολλοί δεν θα χρωστάνε τόσα πολλά σε τόσο λίγους στην Ευρώπη όσον αφορά το μέλλον της Ευρώπης. Σε ευχαριστώ πολύ. Bene, Eh, ευχαριστούμε πολύ τον Υπουργό. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ε, ερωτήσεις ε, και για την προσοχή σας. Next Περνάμε στο επόμενο θέμα. Ελευθεροτυπία και ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης στον κόσμο. Η συγκεκριά μας είναι η Μαρία Σχάκε. Μαρία Σχάκε. Δεύτερη ανταλλαγή απόψε. Έχετε το λόγο. σε ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Θα ήθελα καταρχά να ευχαριστήσω τους κοιόδης ε, εισηγητές για την πολύ ε, καλή συνεργασία Κάναμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων και νομίζω ότι είμαστε κοντά στο στάδιο τη ψήφιση και νομίζω ότι θα στείλουμε ένα πολύ χειρό μήνυμα σε ό,τι αφορά την ελευθεροτυπία και την ελευθερία των μέσων ενημέρωση. Επίση, να ευχαριστήσω τι οργανώσει τη κοινωνία των πολιτών, του δημοσιογράφου και του άλλου φορεί που συμμετείχαν στην διαδικασία αυτή μέσω του διαδικτύου και με άλλου τρόπου. Είναι πολύ επίκαιρη αυτή η έκθεση Γιορτάσαμε πριν από λίγο την ημέρα της ελευθεροτυπίας και μία χρονική συγκυρία όπου η πίεση για την ε, κατάρτιση της ελευθεροτυπίας είναι όλο και μεγαλύτερη. Οι δημοσιογράφοι σε όλο τον κόσμο συχνά είναι προσπίσονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κάποια ε, αριθμητικά στοιχεία το 2012 8 δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν και χιλιάδες άλλοι ε, δέχτηκαν επιθέσει και προ την κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για να διασφαλίσει ε, την ελευθεροτυπία. Θα πρέπει να συνεργαστούμε με τι κυβερνήσει για να του υπενθυμίσουμε τι ευθύνε του, καθώ και με του δημοσιογράφου και την κοινωνία των πολιτών. Δυστυχώ οι κυβερνήσει στι χώρε του τρίτου κόσμου συχνά καταχρώνται του ε, κανόνε, όχι του νόμου, όχι νόμου που έχουν να κάνουν απαραίτητα με την ελευθεροτυπία και τα μέσα ενημέρωση, αλλά που κάνουν κατάχρηση των νόμων των φορολογικών για την δημόσια ασφάλεια για να περιορίσουν την ελευθεροτυπία και να απειλήσουν τους ε, δημοσιογράφους. Ε, μαζί με τους κοιότες εισηγητές ε, αποφασίσαμε να μην θέσουμε το θέμα της ελευθεροτυπίας σε μεμονωμένες χώρες, αλλά σε διάφορα παρατήματα αναφερόμαστε στον ρόλο των ε, ομάδων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που εργάζονται και προσπίσονται την ελευθεροτυπία και αυτά τα παρατήματα τα, τα συνάπτουμε στην έκθεση. Γιατί θέλουμε να καταδείξουμε πόσο σημαντικό είναι να μην υπάρχει πολιτική ανάμειξη στο έργο των δημοσιογράφων, αλλά να διευκολύνονται για να κάνουν το έργο τους με ανεξαρτησία. Τονίζουμε λοιπόν ότι ο τύπος και τα μέσα θα πρέπει να μπορούν να εργάζονται χωρίς πολιτική πίεση και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικά σε ό,τι αφορά τους δημόσιους ε, τους δημόσια μέσα ενημέρωσης, αλλά και φυσικά σε ό,τι αφορά και άλλες επιχειρήσεις ε, που έχουν ε, και φέρουν μεγάλο μερίδιο της ευθύνης. Επίσης αυτό αφορά και το ψηφιακό περιβάλλον όπου ο τύπος, τα μέσα, η πρόσβαση στην πληροφόρηση θα πρέπει να διατηρείται και για την κοινοφελή της ε, λειτουργία. Επίσης τονίζουμε να, την ανάγκη να παταχθεί η ατιμορρησία μετά από απόπειρες καταπίεσης ή απόπειρες επίθεσης προς δημοσιογράφους. Άρα Πρέπει να σας πούμε ότι κοιτάμε και θέματα συνεργασίας για την αρρωγή των ατόμων αυτό. Θα θέλαμε τέλος να τονίσουμε ότι θα πρέπει να συντονιστούν οι γραμμές του προπολογισμού που εφίστανται στο ευρωπαϊκό προπολογισμό και να μην ξεχνάμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παίξει υποδειγματικό ρόλο στο παγκόσμιο προσκήνιο, θα το δώσει το σωστό παράδειγμα Θέλουμε να υπάρχουν ορόσημα σε ό,τι αφορά την επίτευξη των στόχων και να επικεντρωθούμε στην γειτονία μας, στη γειτονιά μας, αλλά να κοιτάξουμε και τις πολιτικές ε, γειτονίας, ε, διεύρυνσης και ούτω καθεξής, προκειμένου να είμαστε πιο αποτελεσματικοί σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση των πόρων σε εποχές περικοπών και ύφεση, προκειμένου να προσπιστούμε αυτέ τι αξίε που είναι τόσο σημαντικέ για μα, την ελευθερία έκφραση, ε, ελεύθερα μέσα ενημέρωση. Όλα αυτά βρίσκονται στον πυρήνα τη ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Και αυτό είναι εν συντομία το περιεχόμενο της έκθεση και προσβλέπω στη μελλοντική μα συνεργασία με τους σκιώδε συζητητέ. Ευχαριστώ πολύ. Δύο ομιλητέ έχω την κυρία Μπρισάτζης πρώτα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά και να συγχαρώ την εισηγήτρια και να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και τους ε, σκιώδης για την καταπληκτική τους προσπάθεια. Καταφέραμε τελικά να συμφωνήσουμε σε όλες τις βαστικές ε, τροπολογίες. Εκ μέρους του ΕΛΚ θα ήθελα να πω ότι θα στηρίξουμε και θα υπερψηφίσουμε όλες τις τροπολογίες, τις συμβαστικές. Έχουμε κάποιες μικρές διαφορές με την εισηγήτρια. Είδα πριν από πέντε λεπτά μόνο τον κατάλογο ψηφοφορίας, αλλά ελπίζω να μείνουμε στην ε, γενική προσέγγιση και να μην χαθούμε σε λεπτομέρειες ή να κατανομάζουμε ε, άτομα ή χώρες. Νομίζω ότι θα έχουμε άλλη ευκαιρία και πιο κατάλληλο θέμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να το κάνουμε και ευχαριστώ θερμά την εισηγήτρια που εστερνίστηκε αυτή την άποψη. Να κρατηθούμε στη γενική προσέγγιση και να μην κατονομάζουμε. Επίσης, ε, το θέμα της, ε, των συντακτών ε, ιστιολογίων, blogger και το θέμα του ίντερνετ δεν το συζητήσαμε αρκετά. Χαίρομαι που το αναβάθμισε η συγγήτρια γιατί είναι πολύ σημαντικό θέμα αυτό. Ιδιαίτερα για κάποια καθεστώτα. Όσο πιο δύσκολο είναι το καθεστώς και πιο φταρχικό τόσο περισσότερο φοβάται ε, το ίντερνετ και τους bloggers, τους συντάκτες των ιστιολογίων. Χαίρομαι λοιπόν που τελικά περιληφθήκε και αυτό το θέμα στην ε, γνωμοδότηση. Θα υπερψηφίσουμε όλες τις συμβαστικές τροπολογίες. Σε μερικά σημεία θα ψηφίσουμε διαφορετικά από την εισηγήτρια βέβαια, αλλά για τεχνικούς περισσότερους, περισσότερο λόγους. Και επειδή έχουμε κάπως διαφορετική πολιτική προσέγγιση από την εισηγήτρια. Αλλά γενικώ είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα και την τροπή των συζητήσεων επί της εκθέσεως. Κύριε Γεκονσάρη, ευχαριστώ και ευχαριστώ την εισηγήτρια την κυρία Σχάκη για την αγαστή συνεργασία που είχαμε και τις πολύ καρποφόρες διαπραγματεύσεις. Χαίρομαι ιδιαίτερως γιατί και εγώ προσωπικά αλλά και και η πολιτική μου ομάδα ικανοποιηθήκαμε γιατί εισακούστηκαν ε, τα αιτήματά μας από την εισηγήτρια στις συμβαστικές τροπολογίες. Οπότε καλύφθηκαν τα βασικά σχόλια των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών που ήταν πρώτα η προστασία των δημοσιογράφων και του έργου τους και η λήψη υπόψη των της ε, αρνητικής πορείας ε, της που έχουν πάρει η ελευθερία του τύπου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Θέλουμε περισσότερο πλουραλιστικό και πολυσχεδί τύπο και ένα πρόσφορο έδαφος και να καταπολεμηθούν κάποιες μονοπολιστικές, μονοπωλιακές συγγνώμη, τάσεις σε ό,τι αφορά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτά ήταν τα αιτήματά μας και συμπεριληφθήκαν. Επίσης, ε, μιλήσαμε για την υποχρέωση της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης να δράσει και να αξιοποιήσει τα εργαλεία και τους μηχανισμούς που έχει σε όλες τις συμφωνίες ε, ε, και συμφωνίες εταιρικής σχέσης ή σύμβαση με τρίτες χώρες. Θα πρέπει το θέμα της ελευθεροτυπίας και της ελευθερίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης να λαμβάνονται υπόψη στις συζητήσεις για τις διάφορες συμφωνίες. Επίσης χρειαζόμαστε μια πιο στενή και διαφανή συνεργασία μεταξύ της ΕΙΕΔ, Τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και να ξαναευχαριστήσω την εισηγήτρια, γιατί η έκθεση έχει λάβει πιο συγκεκριμένη μορφή και περιεχόμενο και δίνει σαφέστερες κατευθύνσεις για μια ενωσιακή στρατηγική. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Να σας υπενθυμίσω ότι η ψηφορία θα λάβει χώρα αύριο στις 5 το απόγευμα. Θέλετε να θέσετε μια ερώτηση. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα μόνο να απαντήσω στα σχόλια τα οποία ακούσαμε από τους κοιόδες συζητητές. Έτσι ε, συντομία, γιατί νομίζω ότι είναι σαφές ότι διακατεχόμεθα από ένα ομαδικό πνεύμα και ότι είναι σημαντικό το θέμα το οποίο πραγματευόμαστε. Θεωρώ λοιπόν ότι η ψηφοφορία θα μας οδηγήσει σε ένα παρόμοιο συμπέρασμα. Θα αποστείλουμε ένα ε, σημαντικό μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση για πολιτικές με καλύτερη στόχευση και με μεγαλύτερη ηγεσία από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά την ελευθερία του τύπου και των μέσων ενημέρωση. Όλοι πιστεύουμε ότι το θέμα αυτό θα πρέπει να είναι στην κορυφή των προτεραιοτήτων μα και ελπίζουμε να υπάρχει πραγματική ε, διαφορά, πραγματικό αποτέλεσμα για τα άτομα αυτά τα οποία διακινδυνεύουν τη ζωή τους και προασπίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και ε, στυλιτεύουν τις αδικίες σε όλο τον κόσμο. Για αυτόν τον κόσμο λοιπόν, για αυτούς τους ανθρώπους γράφουμε την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ πολύ λέει ο Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση αυτή. Περνάμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη για τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την πρόθεση της ευρύτερης διπλωματικής εταιρικής σχέσης. Ο Φρανσίσκο Χωσέ Μιλενμόν είναι ο εισηγητής. Έχετε το λόγο. Ε, Θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω όχι μόνο τον πρόεδρο που μου έδωσε το λόγο, αλλά και τους και οδησηγητές. Οι περισσότεροι απουσιάζουν βέβαια, αλλά και ο κύριος Ρόουτσεκ και η κυρία Νέιτς ε, συνεργάστηκαν μαζί μου πολύ επικοδομητικά. Να ευχαριστήσω τον κύριο Μπουτικόφερτ, γιατί πριν από μια εβδομάδα στο Στρασβούργο συνεννοηθήκαμε και συγκεκριμενοποίησαμε ένα πολύ επικοδομητικό ε, κατάλογο συμβαστικών τροπολογιών. Έχετε λάβει λοιπόν τις συμβαστικές τροπολογίες, οι οποίες καλύπτουν τις μισές τροπολογίες, είτε άμεσα είτε έμεσα. Μπορώ να πω και περισσότερες από τις μισές τροπολογίες, οπότε δεν θα αναφερθώ σε αυτές. Να, να, να πω ότι η έκθεσή μου απαρτίζεται από δύο σκέλη. Το ένα αφορά τι διατλαντικέ σχέσει, τι πιο κλασικέ, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένε Πολιτείε. Και έχω και κάποιου παραγράφου για τι διεθνεί ε, συγκρούσει ε, ή κάποια επίκαιρα ζητήματα, γιατί όλοι επιθυμούμε ε, οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Ευρωπαϊκή Ένωση να δρουν συντονισμένα. Και έχουμε και ένα κεφάλαιο πιο ασυνήθιστο που αφορά μια πιο παγκόσμια διατλαντική προοπτική για το θέμα αυτό υποβλήθηκα λιγότερε τροπολογίε. Ελπίζω να μην οφείλεται αυτό στην αδιαφορία των συναδέλφων για το συγκεκριμένο αντικείμενο. Θα ήθελα τώρα να πω κάτι για τις τροπολογίες. Εγώ θα τις χώριζα στις εξή κατηγορίες. Είναι οι τροπολογίες που συμπληρώνουν, βελτιώνουν ε, ε, την έκθεσή μου και γι' αυτό έβαλα θετικό πρόσημο στον κατάλογο ψηφοφορίας και περισσότερες καλύπτονται και από τις συμβαστικές τροπολογίες. Βέβαια έχουμε κάποιους περιορισμούς στην έκταση, γι' αυτό ε, χάρη στις τροπολογίες εμπλουτίστηκαν και βελτιώθηκαν κάποιες παράγραφοι. Τώρα, άλλες τροπολογίες α, απέκλαιναν από τη βασική γραμμή της έκθεσης, γι' αυτό και έβαλα αρνητικό πρόσημο, αλλά ελάχιστες είναι αυτές. Οι υπόλοιπε τροπολογίες ε, που επίσης θα έχουν ε, αρνητικό πρόσημο είναι εκείνες που διαχωρίζουν τη θέση τους από συγκεκριμένα θέματα της έκθεσης. Για παράδειγμα, όταν έχω μια τροπολογία που δεν θέλει ε, ε, διατελετικό πολιτικό συμβούλιο ή δεν θέλει με τη δεδομένη κατάσταση των δαπανών να κρατήσουμε το γραφείο συνδέσμου το διακοινοβουλευτικό στη Washington, δεν μπορώ να βάλω θετικό πρόσημο σε αυτές τις τροπολογίες που αντιβαίνουν στις δικές μου προτάσεις. Είδα ότι μόλις κατέφτασε και ο κύριος Ρόουτσεκ. Θα, θα το αφήσω λίγο χρόνο να βάλει τα ακουστικά του. Να επαναλάβω τις ευχαριστίες μου για την επικοδομητική μας συνεργασία και να αναφερθώ σε κάποιες άλλες τροπολογίες που εστιάζονται υπερβολικά στο οικονομικό σκέλος του, της εταιρική σχέσης εμπορίου και επενδύσεων, αλλά με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Και το είπα δύο φορές στις συζητήσεις που είχαμε προηγουμένως, ότι θα προσπαθήσω να σεβαστώ τις αρμοδιότητες της ΣΥΝΤΑ και να επικεντρωθώ στα πιο πολιτικά ε, στις πιο πολιτικές και γενικέ πτυχές του TTIP και να μην ε, αναφερθώ σε πιο συγκεκριμένα οικονομικά θέματα που άπτουν τι αρμοδιότητε περισσότερο του ΙΝΤΑ ή κάποιε διαδικαστικέ πτυχέ των διαπραγματεύσεων. Οπότε από αυτήν την άποψη και στι ε, τροπολογίε αυτέ θα βάλω μείον, όχι μόνο για λόγους ουσία, αλλά και για λόγου σκοπιμότητας. Πριν από δύο εβδομάδε η Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου ενέκρινε ένα ψήφισμα συγκεκριμένο για το θέμα αυτό. Πάνω από 22-23 παραγράφου είχε το ψήφισμα αυτό και κάλυπτε ένα το φάσμα και διαδικαστικών και ουσιαστικών θεμάτων που αφορούν τι διαπραγματεύσει. Δεν θα πρέπει λοιπόν να επαναλαμβανόμαστε και να έχουμε μέσα σε δύο μήνε δύο διαφορετικά ψηφίσματα για το ίδιο θέμα. Και θα πρέπει να σεβαστούμε και το διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων. Γι' αυτό και θα βάλω αρνητικό πρόσημο στι τροπολογίε αυτέ που αφορούν είτε διαδικαστικέ είτε ουσιαστικέ πτυχέ των διαπραγματεύσεων. Και έχουμε και άλλε τροπολογίε που δεν θα τι δεχτώ, όχι γιατί δεν μου αρέσει το περιεχόμενο, αλλά γιατί αφορούν πολύ λεπτομεριακά θέματα που ξεφεύγουν από το αντικείμενο της έκθεσης ή που αναλύουν υπερβολικά εξορυχιστικά κάποια ζητήματα. Για παράδειγμα, κάποιες τροπολογίες αφορούν τη συνεργασία για την επιχείρηση Αταλάντη ή για τη Σομαλία. Σε μια γενική έκθεση, όπως η δική μου, που αφορά το Ατλαντικό, αν πρέπει να επεκταθούμε σε ειδικό και ανώ σε ειρηνικό, νομίζω ότι παραπάει. Too much, όπως λέμε και στα αγγλικά. Είναι υπερβολικό. Το παρατραβάει θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για τον κόλπο του Άντεν, για τον ε, κόλπο του Άντεν, για την Αταλάντη, για τη Σομαλία, για τον Ειδικό. Δεν μπορούμε να τα λέμε όλα. Για τι ατλαντικές σχέσει μιλάμε. Γι' αυτό θα βάλω αρνητικό πρόσημο. Ούτε υπερβολικέ λεπτομέρειε έχουν θέση στην έκθεση. Δεν έχουμε έκθεση εδώ για την ενευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, ούτε για τι κλιματικέ αλλαγέ, ούτε για ενεργειακά ζητήματα, ούτε για τον ΝΑΤΟ. Οπότε τέτοιε τροπολογίε που ξεφεύγουν από το αντικείμενο τη έκθεση που διευρύνουν υπερβολικά το περιεχόμενο θα λάβουν αρνητικό πρόσημο. Επίσης, στην προηγούμενη συζήτηση η κυρία Νέιτς και ο κύριος Μπιουτικόφερ μου προσήψαν ακριβώ ότι στην έκθεσή μου δεν επικεντρωνόμουν σε συγκεκριμένε προτεραιότητε και ότι επεκτηνόμουν σε πολλά θέματα. Το έλαβα υπόψη λοιπόν αυτή την φιλική μορφή και προσπάθησα να περιορίσω αυτή την έκθεση, να μην ε, το κάνουμε υπερβολικά στολισμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο, γιατί αλλιώς θα, θα γινόταν ε, ένας ε, χήμαρος αυτή η έκθεση που θα κατέκλυζε τα πάντα. Επίσης, πρόκειται για μια έκθεση που στρέφεται προς το μέλλον. Δεν επικεντρώνεται στο παρόν ούτε στο παρελθόν. Βρισκόμαστε ήδη στο δεύτερη θητεία του Ομπάμα. Περάσαμε το, τη φάση Μπούς. Διανύουμε μια περίπλοκη και σύνθετη, σύνθετη περισσότερο θα έλεγα παρά περίπλοκη και δύσκολη σχέση με τη ΣΥΠΑ. Έχουμε την, ε, το, το Leading for Behind, το δόγμα, έχουμε την ε, αναδυόμενη Ασία, έχουμε διάφορες κρίσεις, την επανάληψη των α, ε, διατλαντικών διαπραγματεύσεων για το εμπόριο και τις επενδύσεις. Ας αφήσουμε λοιπόν το παρελθόν και ας στραφούμε προς το μέλλον. Οπότε οι τροπολογίες που παρελθοντολογούν κάπως δεν θα με βρουν σύμφωνο. Για να μην σας κουράσω λοιπόν θα ολοκληρώσω λέγοντα ότι και η έκθεσή μου αλλά και οι συμβαστικέ τροπολογίε και ο κατάλογος ψηφοφορία στόχο έχουν να διαμορφώσουν μια ισορροπημένη έκθεση, φιλόδοξη, περιεκτική, αλλά με κάποιες προτεραιότητες. Δεν μπόρεσα να τα συμπεριλάβω όλα, λογικό ήταν. Πάντως όσοι είχαν την υπομονή να ακούσουν μέχρι το τέλο, θα λάβουν το λόγο και περιμένω και εγώ με ιδιαίτερη ανυπομονησία να του ακούσω και να ακούσω και τι προτάσει του. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχά να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εξαιρετική του δουλειά, για την ε, επικοδομητική συνεργασία, για την έκθεση. 22 τροπολογίες ε, προέκυψαν και νομίζω ότι στις συμβαστικές προτάσεις περιλαμβάνονται και οι τροπολογίες των σοσιαλδημοκρατών αλλά και των άλλων ομάδων από πλευρά της ομάδα μου να σας πω ότι μπορούμε να τις υποστηρίξουμε όλες τις συμβαστικές προτάσεις. Το τελικό αποτέλεσμα νομίζω ότι είναι στεναρό και επιβεβαιώνει εκ νέου την δέσμευση του Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά την υποστήριξη των διακρατικών σχέσεων και επίσης θεωρώ ότι διατυπώνει κάποιες ιδέες οι οποίες θα πρέπει να προαχθούν αλλά και κάποιες καινούργιες ιδέες. Είναι λοιπόν επίκαιρη ε, σχετική με το τρέχον αντικείμενο η έκθεση, καταστά σαφές ε, το αντικείμενο των διακλαντικών σχέσεων που βρίσκονται σε περίοδο μεταβολής ε, λόγω της οικονομικής κρίσης, λόγω των αναδυόμενων δυνάμεων στην Νοτιοανατολική Ασία και φυσικά περιλαμβάνονται και ζητήματα που αφορούν την Αραβική Άνοιξη. Αναφέρεται λοιπόν η πτυχή της ε, πιο στενή συνεργασία και τη πιο στεναρή ε, διαδικατικής σχέση. Αναφέρεται η διαδικασία τη DIP, η οποία είναι πολλά υποσχόμενη, όχι μόνο σε ό,τι αφορά το οικονομικό το όφελος, αλλά και το γεωπολιτικό όφελος. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε την ορμή αυτή για την ε, προώθηση των διατρατικών σχέσεων και σε ό,τι αφορά και την εξωτερική πολιτική. Όπως είπε όμως ήδη ο εισηγητής, η Επιτροπή ΙΝΤΑ αποτελεί την καθήλια αρμόδια Επιτροπή για την διαπραγμάτευση της TTIP. Δεν πρόκειται λοιπόν να μπούμε στα δικά τους χωράφια. Σύμφωνο λοιπόν μαζί του για το γεγονός ότι δεν υποστηρίζει κάποιες από τις τροπολογίες επειδή επισέρχονται στα νερά της Επιτροπής ΣΥΝΤΑ. Θεωρώ επίσης ότι βλέπουμε με σαφήνεια να διαμορφώνεται ένα πλαίσιο για μία ευρύτερη ε, σχέση, διδελτική σχέση. Να μην ξεχνάμε τον Καναδά, να μην ξεχνάμε νέες δυνάμεις στη Λατινική Αμερική, να μην ξεχνάμε αφρικανικές δυνάμεις που θα ήθελαν ενδεχομένω να συμμετάσχουν με κάποια μορφή στην διατλαντική ατζέντα. Αναφέρονται όλα αυτά στην έκθεση. Χωρίς ωστόσο να υπονομεύουν την πιο στενή σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΠΑ. Να συγχαρώ λοιπόν τον κύριο Μιλανμόν να τον ευχαριστήσω για το επικοδομητικό του πνεύμα και προσβλέπω στην αυριανή ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Σάκε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφε μιλανμον μιλώ εξ ονόματος της κυρίας Νέιτς, η οποία ζητά συγγνώμη γιατί δεν μπόρεσε να μείνει με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολούθησα την εξέλιξη της έκθεσης, η οποία θεωρώ ότι είναι αρκετά ευρία στο πεδίο εφαρμογής της, αλλά και πάλι αποτυπώνει σωστά εικόνες, σωστές ε, ιδέες για την τελική σχέση. Σας ευχαριστώ λοιπόν η ομάδα μας για το έργο σας ως μέλος της Επιτροπής ε, Διεθνούς Εμπορίου. Ασπάζομαι την άποψή σας για το ότι δεν ε, χρειάζονται επικαλύψεις είναι σημαντικό το έργο που έχει να κάνει και η Επιτροπή Εκτορικών Υποθέσεων αλλά και η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου όπου πρόσφατα υπερψηφίστηκε μια έκθεση η οποία θα διαμορφώνει την σχετική διαπραγματευτική εντολή για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συμφωνούμε με το όραμά σα για το μέλλον τη διευθυντική σχέση. Είναι σημαντικό να υπάρχει σημασία σε μια τέτοια εποχή μεταβολών και αλλαγών και εξετάζοντας τον κόσμο αυτόν όπως αλλάζει, είναι σαφές ότι η δέσμευση της επόμενης γενιά για την διατελική σχέση δεν είναι κάτι δεδομένο. Θα χρειαστεί ηγεσία από πλευρά μα για να δοθεί νέο μήνυμα, νέα ουσία και από πλευρά οικονομική. Και νομίζω ότι αυτά αποτυπώνονται πολύ σωστά στην έκθεση και από πλευρά γεωπολιτική και από πλευρά υπογράμμιση τη ανάγκη για στενατορή συνεργασία και για οικονομικούς, επενδυτικούς, εμπορικούς δεσμούς. Αυτές οι προσθήκες λοιπόν είναι καλές και θεωρώ ότι θα διαμορφώσουν μέσα στον τρόπο το μέλλον της διακρατικής σχέσης. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος, να κάνω και εγώ κάποιες παρατηρήσεις, να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Μίλαν Μόν για την έκθεση αυτή που προχωρά τις διατλαντικές σχέσεις. αναφέρεται και στις ε, διαπραγματεύσεις που ξεκινούν για την διαδικατική αγορά και στη σημαντική πολιτική διάσταση και στις εμπορικές συνέπειες. Μία ερώτηση να κάνω και εγώ στους συναδέλφους. Οι συστάσεις της ε, Επιτροπής ε, Διεθνούς Εμπορίου θα ψηφιστούν στην Ολομέλεια το Μάιο, ενώ η έκθεση του συναδέλφου Μίλαν Μόντ θα ψηφιστεί τον Ιούνιο. Δεν θα ήταν καλό να γίνει μια συζήτηση από κοινού. Ίσως θα έπρεπε οι συντονιστέ να το ζητήσουν να υποβάλουν σχετική αίτηση, γιατί αν αύριο υπερψηφίσουμε την έκθεση, έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίε να, να διαμοιραστεί στις ε, ομάδες και να τη συζητήσουμε στο Στρασβούργο. Ίσως θα μπορούσαν λοιπόν να το σκεφτούν αυτό οι ομάδες. Μου φαίνεται πιο λογικό τι να σας πω. Να τα συζητήσουμε από κοινού. Ίσως θα μπορούσαν να το συζητήσεις και με τον συναδελφό Μονέρα για να μην ε, παρουσιάσετε τις συνήθεις δυσκολίες. Κύριε Πρόεδρε, οι διαδηλατικές σχέσεις διανύουν μια συγκεκριμένη πολύ ιδιαίτερη στιγμή όπως ένα των διαπραγματεύσεων, αλλά πέραν τούτου υπάρχουν και άλλα θέματα. Και αυτή η έκθεση δεν επικεντρώνεται μόνο στην κλασική διατλαντική σχέση, αλλά έχει ευρύτερο περιεχόμενο. Μίλησε για το Νότιο Ατλαντικό. Και από αυτήν την άποψη είναι καινοτόμα η έκθεση. Περιλαμβάνει και τη Λατινική Αμερική και τη Δυτική Όχθη της Αφρικής. Και ναι, μένει στις 18, 19 ή 20 Ιουνίου έχουμε ε, G8 και ο πρόεδρος Ομπάμα θα έρθει 17-18 στη Βόρεια Ιρλανδία. Οπότε αν εμείς εγκρίνουμε την έκθεση 14, 15, 16 Ιουνίου, αν τότε την συζητήσουμε και την ε, εγκρίνουμε, άσχετα με το ψήφισμα της ΣΥΝΤΑ που θα πάει το Μάιο, οπότε αν η δική μας έκθεση εγκριθεί 3-4 μέρες πριν την ε, άφηξη του Ομπάμα στην Ευρώπη είναι πολύ επίκαιρο νομίζω και δεν είναι άμερο σημασία. Και δεν είναι κακό ή ανόητο να διαχωρίζουμε τις δύο εκθέσεις. Οπότε αν η συζήτηση γίνει ε, και για τις ε, δύο εκθέσεις, δεν ξέρω αν από τη δικαστική άποψη είμαστε εντάξει με τις τροπολογίες και τις ε, ψηφοφορίες. Έχουμε πρώτα την αυριανή ψηφοφορία, αλλά δεν θα πρέπει να επισκιάζεται η έκθεσή μας από την έμφαση που θα δοθεί μόνο στα οικονομικά και εμπορικά θέματα. Ενώ αν την αφήσουμε για τον Ιούνιο, μπορεί να έχει προηγηθεί ψηφοφορία της ΣΥΝΤΑ, αλλά η δική μας θα ψηφιστεί τρεις-τέσσερις μέρες πριν την αύξηση των Ομπάμα στην Ευρώπη και τη διμερή διάσκεψη κορυφής. Και όλοι ξέρουμε ότι θα έχουμε τη διαπραγματεύσεις για, τη, για το διατλαντικό εμπόριο, αλλά η έκθεση μου είναι ευρύτερη. Οπότε δεν είναι άσκοπο κατά τη γνώμη μου η παράλογο να το αφήσουμε για τον Ιούνιο. Σκέφτομαι μέχρι αύριο, για όλα υπάρχει κάποια, κάποιος λόγος. Τρεις πριν από το ταξίδι του Ομπάμα. Ναι, θα πρέπει να έχουμε αποφασίσει γιατί αλλιώ δεν θα περιλαμβάνονται αυτά στα χαρτιά του Ομπάμα. Λίγο φοβάμαι για θέματα διαπραγματευτικά όταν ε, γίνουν καθαρά εμπορικά ζητήματα, εμπορικά ζητήματα θα χάσουμε την ορμή. Γιατί αυτές οι διαπραγματεύσεις έχουν και ε, μια διάσταση πολιτικής ασφαλείας. Γι' αυτό λοιπόν για πολιτικούς λόγους θα ήθελα να τα κοιτάξουμε αυτά από κοινού και όχι να τα διαχωρίσουμε, να το σκεφτούμε. Και να δούμε κατά πόσον τεχνικός πώς ε, προλαβαίνουμε και για τις μεταφράσεις και για τα υπόλοιπα. Sí, señor presidente, muchas gracias. Yo creo que el criterio fundamental a la hora de tomar una decisión. Νομίζω το σημαντικότερο κριτήριο για να ληφθεί μια απόφαση για το πότε θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση είναι ότι πρέπει κανείς ε, να λάβει υπόψη τα υπέρ και τα κατά και αυτό να το αποφασίσει ο εισηγητής. Μετά την ε, ψηφοφορία θα πρέπει να έχουμε χρόνο να εξετάσουμε τα υπέρ και τα κατά. Αν όλα αυτά θα τα ε, συνδυάσουμε με τα εμπορικά θέματα και με το όταν θα έρθει ο πρόεδρος Ομπάμα στην Ευρώπη. Νομίζω λοιπόν ότι η απόφαση είναι καλύτερα να ληφθεί από τον εισηγητή, ίσως από κοινού με τους ε, σκιώδη εισηγητέ, γιατί πράγματι η δουλειά που έχει γίνει στην έκθεση αυτή είναι πάρα πολύ καλή. Πρέπει μετά την ψηφορία να τους δείξουμε εμπιστοσύνη και να αποφασίζουν μόνοι τους το πώς θα προχωρήσουμε. Εντάξει, λέει ο Πρόεδρος, θα το συζητήσουμε αύριο, γιατί αύριο πρέπει να ληφθεί η απόφαση αύριο είναι και η διορία. αλλιώ και καθαρά τεχνικά πλέον δεν γίνεται τίποτα. Ίσως και σήμερα το βράδυ να μπορέσουμε να μιλήσουμε λιγάκι για το θέμα αυτό. Πάντως ε, δεν επιθυμώ το θέμα αυτό να μην εξεταστεί ε, στην Επιτροπή μας και εμείς να είμαστε ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Δεν μ' αρέσει αυτό. Λοιπόν, τελειώσαμε. Αύριο το πρωί στις 5 ώρα είναι η ψηφοφορία. Γεια σας.